Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Our program for today is very busy. Είναι κατάμεστη η μερίσια μας διάταξη σήμερα και το πρόγραμμά μας πλήρες. Γι' αυτό παρακαλώ και, έχουμε ήδη καθυστερήσει ένα δεκάλεπτο. Καθίστε για να ξεκινήσουμε αμέσως. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν σχόλια ή προτάσεις για την ημερήσια διάταξη? Όχι, οπότε μπορούμε να την εγκρίνουμε. Σημείο 2. Έγκριση των σχεδίων πρακτικών των συνεδριάσεων της 20ης Ιουνίου, 25ης Ιουνίου και 10ης Ιουλίου 2018. Τα πρακτικά υπάρχουν στο διαδίκτυο, οπότε ο συνήθως αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μέχρι το τέλος συνεδρίασης, θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Δεν βλέπω άλλα σχόλια και προχωρώ. Σημείο 3. Ανακοινώσει τη Πρόεδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Απλώ να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που σα ξαναβλέπω όλου εδώ σήμερα και ελπίζω να περάσετε καλά το καλοκαίρι στι διακοπέ σα. Να απολαύσετε το καλοκαίρι είτε στην πατρίδα σας είτε σε ταξίδια και να είστε ακμαίοι και να σφίζετε από ενέργεια ώστε να ανταποκριθούμε στο απαιτητικό έργο τους επόμενους μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν η μόνη ανακοίνωση που είχα. Και προχωρούμε στον ε, ε κανονισμό 1303 του 2013 που αφορά τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη διόρθωση του κανονισμού που αφορά τους πόρους ε, για τις επενδύσεις ε, στους στόχους της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στις 28 Ιουνίου τρέχοντος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα νέο, μια νέα πρόταση για την τροποποίηση του εφιστάμενου μηχανισμού, ε, κανονισμού κοινών διατάξεων με δύο σημεία. Καταρχήν, μερικά κονδύλια και πιστώσεις του 2020 μεταφέρονται στο 2018 για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Αυτό συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2018. Και μάλιστα η αύξηση είναι σημαντική, 116,7 εκατομμύρια, κάτι που φέρνει τον συνολικό προπολογισμό για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων για το 2018 στα 350 εκατομμύρια. Δεύτερη πρόταση, διορθώνονται κάποια στοιχεία του άρθρου 92 παράγραφος 1 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, ε, γιατί κάποια στοιχεία του αναθεωρημένου κανονισμού ήταν ανακριβή. Ως εισηγήτρια, η Πρόεδρος προτείνει να υπαχθεί αυτή η διαδικασία στο ο κανονισμός στη διαδικασία του άρθρου 50 παράγραφος 1 να εγκριθεί δηλαδή με την απλουστευμένη διαδικασία και χωρίς τροπολογίες. Ήδη σας έχουμε μοιράσει με τα έγγραφα της συνεδρίασης στο σχέδιο έκθεσης της ε, Προέδρου και ρωτώ αν υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς τη χρήση της απλουστευμένης διαδικασίας για την έγκριση του κανονισμού. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Σας ευχαριστώ. Τέστην Εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες. Δεν χρειάζεται καν να ψηφίσουμε για το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε αυτή την εξαίρεση και την επαγωγή στην απλουστευμένη διαδικασία. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Αφού δεν έχουμε άλλα σχόλια, να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Να βγάλω και την κάρτα μου. Ξεκινούμε με την ψηφοφορία για το Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοσιονομική Χρήση του 2019. Όλα τα τμήματα. Πρόκειται για γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα με συντάκτη τη γνωμοδότηση τον κύριο Ντέρεκ Βον. Θα ήθελατε το λόγο, έχετε να πείτε κάτι κύριε Σιγητά. Όχι, οπότε να πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Έχουμε και συμβαστικές τροπολογίες. Ξεκινάμε με τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε πανψηφή. Συγχαρητήρια κύριε Βόν. Okay. Uh, the second Περνάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία για την αύξηση του κονδυλίου για το πρόγραμμα στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσαρμογή του γενικού του στόχου. Υπό την καθοδήγηση τη ηγέτριά μα, τη κυρία Ρούζα Τόμασιτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη διαπραγματευτική ομάδα κατέληξε συμφωνία στον τριμερή διάλογο τη 11η Ιουλίου ως προς την πρόταση αναθεώρηση του κανονισμού 2017 κάθετος 825 για την αύξηση του κονδυλίου ε, για το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την προσαρμογή του γενικού του στόχου. Το κείμενο της συμφωνίας έχει μοιραστεί, έχει αποστέλει ηλεκτρονικά μαζί με τα έγγραφα της συνεδρίασης στα μέλη της Επιτροπής και θέλει το λόγο η συγκεκριά μας, η κυρία Τόμασιτς, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας σε ό,τι αφορά αυτή την κατεπίγουσα έκθεση. Έχω επίγνωση του τεχνικού χαρακτήρα της, γιατί οι αλλαγές είναι λίγες και ανεπαίσθητες. Παρ' όλα αυτά, ε, θα ήθελα να είχαμε περισσότερο χρόνο για να περιλάβουμε όλες τις αλλαγές. Η διορία για τα κράτη-μέλη για να υποβάλουν τις προτάσεις της, είναι τέλειο Οκτωβρίου, τρέχοντος έτους για τις προτάσει για το SRSP για το 2019 και ελπίζω να εγκριθούν σήμερα οι σχετικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε άπαξ, γιατί δεν μπορούμε παρά να εγκρίνουμε να απορρίψουμε την πρόταση και θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Η έκθεση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Τόμασιτς. Ωραία, ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και περνάμε στο σημείο 7 θα συζητήσουμε τις νέες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και η πρώτη συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει σήμερα χάρη στον κύριο Αριμό με θέμα τις ειδικές διατάξεις για το στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των εξωτερικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στις 29 Μαΐου τρέχοντος έτους λάβαμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κύριος Αριμόν ανέλαβε την έκθεση εκ μέρους της Επιτροπής μας για το Interreg. Σήμερα ο κύριος Αριμών θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα το χρονοδιάγραμμα υπό το, υπό το οποίο συντάχθηκε η έκθεση αρχές Ιουλίου ορίστηκα εισηγητής. Πρώτο συζητήσαμε την έκθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχές Ιουλίου έγραψα το κείμενο τις τελευταίες δύο εβδομάδες του Ιουλίου και το συνέταξα με τρόπο ώστε να μας επιτρέπει σε εμά ως Επιτροπή να περιλάβουμε και τις απόψεις των συναδέλφων. Αυτό είναι ο σκοπός τώρα με την κατάθεση τροπολογιών. Είναι η πρώτη συζήτηση σήμερα της έκθεσης. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω πίεσης χρόνου εργαστήκαμε ταχύτατα μπορέσαμε να συναντήσουμε ορισμένους από τους βασικούς ενδιαφερομένους φορείς, αλλά όχι όλους γιατί ήταν και οι διακοπές. Όλα αυτά τα περιλάβαμε στην έκθεση. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι διατηρεί το στοιχείο της εδαφικής συνοχής και τα προγράμματα τα συνεχίζει. Τα λέω αυτά διότι είμαι σαφώς υπέρ του προγράμματος Interreg. Άλλωστε προέρχομαι από μια περιοχή σε τριεθνή σύνορα και αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ποιε είναι οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που κατοικούν σε μια χώρα και εργάζονται σε κάποια άλλη. Γι' αυτό και επιθυμώ να υποστηρίξω τα προγράμματα αυτά, διότι μα επιτρέπουν να επιτύχουμε πολλά πράγματα, Ιδίω στι σημερινέ συνθήκε που ζούμε στην Ευρώπη, και όπου η Ευρώπη, ίσως η ιδέα της Ευρώπης, ε, την ιδέα μάλλον της Ευρώπης, είμαστε υποχρεωμένοι να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι υπερεθνικές συνεργασίες που επιτρέπουν σε ανθρώπους να συνέρχονται, να αναζητούν λύσει από κοινού, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη διαφήμιση που μπορούμε να κάνουμε υπέρ τη Ευρώπη στι σημερινέ συνθήκε. Θα ήταν αμέλεια εκ μέρου μα εάν διαγράφαμε το ίντερνετ ή απλώ και το περικόπταμε. Αυτά ως εισαγωγή, διότι αυτές οι περιφέρειες γίνονται τελικώς πολύ σημαντικά στοιχεία για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε το, τους σκοπούς αυτούς. Σας λέγω με λίγα λόγια τι τροποποιώ στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσα να σας πω πολλά και για τα όσα δεν τροποποιώ. Θα έρθω κυρίω όμως σε αυτά τα οποία επιθυμώ να τροποποιήσω και πρώτο και βασικό στοιχείο είναι το πεδίο εφαρμογής. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί στις παραμεθόριες περιφέρειες ένας ρόλος κλειδί και πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον και η θαλάσσια ή διαθαλάσσια συνεργασία. που είναι αναπόσπαστο μέρο τη ανάπτυξη αυτή. Εδώ και καιρό λειτουργεί καλά το Interreg. Διερωτώ με λοιπόν γιατί πρέπει άραγε να τροποποιηθεί εφόσον αποδείχθηκε ότι λειτουργεί καλά. Ανοίγουμε τότε έναν ασκό που δεν γνωρίζουμε που θα ε, καταλήξουμε όταν θα τον ανοίξουμε. Γι' αυτό η θαλάσσια συνεργασία πρέπει να μπει στο πρώτο τμήμα του νομοθετήματος και έχω κάνει σχετική τροποποίηση. Υπάρχουν επίσης και ή περιφερειακές επενδύσεις. Αρκετά περίπλοκη διατύπωση και πρόκειται για το τμήμα 5. Εδώ υπάρχουν υπέρ και κατά. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να παραμείνει το Interreg στα όσα ήδη κάνει. Στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, αποκεντρωμένα Αυτά όμως δεν ανεβρίσκονται πάλι στο υπαριθμό 5 τμήμα. Είμαι διατεθειμένος να συζητήσω για αυτό το τμήμα 5, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται να οδηγήσει, να επιβαρύνει δηλαδή τα άλλα. Έρχομαι τώρα στην εγγραφή στον προϋπολογισμό. Τα τμήματα 1 έως 4 θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με τον κατάλληλο τρόπο και ενδεχομένως να αυξηθεί μάλιστα ο προϋπολογισμός τους. Έχω περιλάβει συγκεκριμένα ποσοστά και όταν κάνει κανείς το συνολικό υπολογισμό καταλήγει σε αύξηση του συνολικού ποσού, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται εγώ να το εγγράψω στην έκθεση αυτή, το μόνο που με επιτρέπεται είναι να περιλάβω ποσοστά. Όποιος δεν λαμβάνεται τα ποσοστά όμως αντιλαμβάνεται ότι σιωπηρά νοείται ότι θα υπάρξει τελικά αύξηση του προϋπολογισμού. Εάν οι χώρες μέλη θέλουν πράγματι το τμήμα αυτό 5 ως τμήμα το οποίο θα το ελέγχει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθύτερα στην τσέπη. Σημαντικό για μας, για μένα δηλαδή και για πολλούς που ασχολούνται με τα Interreg προγράμματα επιτόπου, δεν είναι μόνο τα μεγάλα προγράμματα Interreg, αλλά και τα πολλά μικρά ή πολύ μικρά προγράμματα. People to people τα λένε αυτά στα αγγλικά. Όπου για παράδειγμα διοργανώνει μια εορταστική εκδήλωση ένα σύλλογο που έχει μέλη από τρεις διαφορετικές χώρες. Αυτά τα πράγματα βοηθούν διότι δείχνουν ότι η, εικόνα, η, μάλλον η Ευρώπη εγκύπτει στα προβλήματα αυτά τα μικρά και καθημερινά. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο να δώσει μια νομική βάση σε αυτά τα people-to-people projects και το πράττει αυτό στο νέο νομοθέτημα. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 70%. Εμείς το επαναφέρουμε στο 85% όπως ήταν παλαιότερα. Και θεωρούμε επίσης ότι αυτή η συγχρηματοδότηση, οι συντελεστές συγχρηματοδοτήσεως θα πρέπει να είναι εύκαμπτοι, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσει των διαφόρων προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά την προχρηματοδότηση, εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερα αξία στο γεγονός ότι πολλοί που εκτελούν προγράμματα μας είπαν ότι η αρχική φάση είναι και η δύσκολη. Δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη προχρηματοδότηση στην αρχή από ό,τι προς το τέλος. Και γι' αυτό έχουμε αυξήσει τα σχετικά ποσοστά. Στην έκθεσή μου δεν περιλαμβάνω τροποποίηση για το 6% για τη χρηματοδότηση των δομών αυτών, για τον απλό λόγο ότι εκπίπτει ένα επίπεδο λογιστικού ελέγχου, το οποίο μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα δαπανηρό, διότι γινόταν από εξωτερικές εταιρείες ή μπορούσε να γίνεται από εξωτερικέ εταιρείε και ήταν επομένω, επαναλαμβάνω, δαπανηρό. Τα χρήματα που εξοικονομούνται μπορούν να χρηματοδοτήσουν τι δομέ αυτέ. Ευχαρίστω όμω θα το συζητήσω το θέμα αυτό μαζί σα. Από το νη 2 έκανα εγώ, το φτιάξα πάλι νη 3 για να αποφευθεί η απώλεια κονδυλίων και κάτι άλλο οι ρυθμίσεις των επιχορηγήσεων, που είναι και νομικά δύσκολο θέμα, διότι εάν αλλάξουμε κάτι εδώ μπορεί να αποτελέσουν οι αλλαγές αυτές προηγούμενο και αυτό πρέπει να αποφυθεί για προγράμματα, για έργα δηλαδή Interreg το οικονομικό μέγεθος είναι πολύ σχετικό και εν πάση περιπτώσει έχει λίγη επιρροή στο σύνολο της οικονομικής απόδοσης ώστε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι έλεγχοι των επιδοτήσεων μπορούν και να εξαιρεθούν ή εν πάση περιπτώσει να υπάρξει κάποια εξαίρεση ώστε και οι επιτόπου ενδιαφερόμενοι να αποφύγουν τα προβλήματα αυτά διότι ε, χρειάζεται κάθε φορά να αναζητήσουν τη συμβολή δικηγόρου, να δουν δηλαδή εμπίπτουν στις σχετικές ε, ρυθμίσεις ή όχι τα προγράμματα που επιθυμούν να προωθήσουν και το καθεξής και αυτό είναι και χρονοβόρο και δαπανηρό. Εν Θέλω να πω, μιλώντας για τις τροπολογίες, ότι βεβαίως αυτές οι τροπολογίες που έχω καταθέσει δεν είναι και, και ε, σκαλισμένες σε λίθο, ε, μπορούμε να τις αλλάξουμε, τις έκανα από κάποια πίεση χρόνου. Ελπίζω να μπορέσουν να υποστηριχθούν από όσο δυνατόν περισσότερου συναδέλφου, ώστε να είναι ενωμένη και δυνατή η φωνή μα απέναντι στο Συμβούλιο, ώστε το Ίντερεγ να παραμείνει Ίντερεγ και να χρηματοδοτηθεί επαρκώ. το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή η προθεσμία μέχρι την οποία μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες, είναι μόλις η 10η Σεπτεμβρίου. Εάν αυτό αποτελεί πρόβλημα, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να αναστείλουμε την προθεσμία αυτή για τρεις-τέσσερις ημέρες, χωρίς να αλλάξουμε ολόκληρη την ατζέντα όμως, γιατί θα ήταν σωστό και σκόπιμο νομίζω να μπορέσει να ολοκληρωθεί η πορεία της εκθέσεως και του νομοθετήματος επομένως μέσα στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση και ευχαριστώ να λάβω υπόψη όλες τις ιδέες που θα θέσετε υπόψη μου και σήμερα και τις επόμενες ημέρες και να τις περιλάβω σε νέες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ κύριε Αριμόν. Τώρα θα δώσω τον λόγο στους πιο δυσίτες. Έχουμε και την εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιφερειών που έχει αναλάβει γνωμοδότηση για, την, για το ίδιο θέμα, την κυρία Μον Περτό. Θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να της δώσω τον λόγο επίσης. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από την σωστή τήρηση των χρονικών ορίων παρεμβάσεων δικών σας. Σας υπενθυμίζω εξάλλου ότι εδώ ισχύει το άρθρο 54 σε συνεργασία δηλαδή με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Οι εισηγητές των οποίων επιτροπών έχουν προσκληθεί σήμερα να παρευρεθούν στη δική μας συνεδρίαση. Αρχίζω λοιπόν τώρα με τους κοιόδης εισηγητές και στο τέλος θα συζητήσουμε πάλι τις προθεσμίες των τροπολογιών. Ίσως μπορέσουμε να την αναβάλουμε μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, αντί τις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως το τέλος της συζητήσεως. Πρώτα λοιπόν το λόγο να λάβουν οι σκιώδεις συγητές και σας παρακαλώ όλες και όλους να μην υπερβείτε τα τρία λεπτά. Εάν μπορείτε. Καλά, να προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, αν και ίσως είναι κάπως ασύνηθες, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Αριμών για το σχέδιο που έχει συντάξει. Είναι καλό το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει πολλές θετικές ιδέες. Η αντίδραση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε άλλωστε καταρχήν θετική έχει πράγματι μεγάλη σημασία αυτή η απλούστευση που προσπαθεί να προωθήσει. Υπάρχουν βέβαια και κάποια ζητήματα κριτικής και συμφωνώ κύριε ε, Αρημόν ότι όχι μόνο παρακολουθήσατε τι είπαμε, ακούσατε καλά και δράσατε σωστά. Μιλήσατε πριν για τον προϋπολογισμό το ίντερνετ είναι το πρόγραμμα εκείνο το οποίο φέρνει του ανθρώπου κοντά και όπου οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται με ποιον τρόπο ε, διαμορφώνεται η προστιθέμενη αξία τη Ευρώπη. Θα ήταν μοιραίο λάθο να περικόψουμε τον προπολογισμό του Ιντερνετ. Δεν μου επιτρέπεται να το αφήσουμε να γίνει αυτό. Δηλαδή η Ευρώπη δεν πρόκειται να αποδείξει την αξία τη διαπανώντα λιγότερα χρήματα, τουλάχιστον διατηρώντα τον ίδιο προπολογισμό ωστόσο. Ε, συμφωνώ απόλυτα λοιπόν μαζί σου αγαπητέ Αριμών, όπω είπε και εσύ, η μετατόπιση της ε, θαλάσσιας συνεργασίας στο τμήμα 2 δεν έχει κανένα νόημα, ούτε και μου το εξηγήσει κανείς ποτέ αυτό, γιατί θα έπρεπε να γίνει άλλα γι' αυτό. Θα ήθελα να, να διατηρηθούν μάλλον οι δομές ως έχουν. Έχει ενδιαφέρον, το είπε και εσύ προηγουμένως αγαπητέ Αριμών, η η διαπεριφερειακή επένδυση καινοτομία. Είναι μια Ενδιαφέρουσα υπόθεση. Βεβαίω πρόκειται για έναν κάπω περίεργο όρο, αλλά υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τη διαχείριση. Είναι όμω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όμω, γιατί τώρα καινούριο project το οποίο να χρηματοδοτεί με ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το καλάθι του Interreg. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με λιγότερα χρήματα, αλλά νέα χρήματα, όχι από το καλάθι του Interreg. Για το δίκαιο των επιχορηγήσεων, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπες. Όπου και να πηγαίνω μου θέτουν το ίδιο ερώτημα. Για, τα, για το Ταμείο για τα πολύ μικρά project. Το έχω ξαναπεί και εγώ. Είναι και αυτό πάρα πολύ σπουδαίο εργαλείο και να διατηρηθεί. Το ίδιο άλλωστε όπως και εσύ αγαπητέ κύριε Σιγητά υποστηρίζω αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο κάποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Για παράδειγμα πρόγραμμα Pro-Interreg και βεβαίω ε, να μην γίνονται πάντοτε αναγκαστικά πράγματα μέσω νομικού προσώπου. Για την συγχρηματοδότηση, και εδώ νομίζω είναι σωστά αυτά που λες, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό συντελεστή της συγχρηματοδότησης πέραν των προτάσεων αυτών που κάνεις εσύ και ως ό,τι αφορά τον έλεγχο πρώτου επίπεδου νομίζω πρέπει να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες υποβολής εκθέσεων. Εγώ θα κάνω σχετικές τροπολογίες και εξ ονόματος της πολιτικής μου Για την τεχνική βοήθεια, μέχρι τώρα αυτή δεν είχε συζητηθεί καθόλου. Και εδώ λοιπόν θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον και να τις περιλάβω σε εχθρικέ τροπολογίε. Για παράδειγμα, το συνολικό επιτρεπόμενο ποσοστό σφάλματος μπορεί να αυξηθεί, διότι γνωρίζουμε και από το παρελθόν ότι έχουν προκληθεί δυσκολίε εκεί. Μπορούμε λοιπόν να φανούμε λίγο πιο γενναιόδοροι εκεί. Ένα ερώτημα τέλο να μου επιτρέψετε, διότι δεν γνωρίζω ακριβώς πώς πρέπει να το εκλάβω. Σε έναν από τους ειδικού στόχους Ίντερεκ λέει μεγαλύτερη ασφάλεια για την Ευρώπη. Το ερώτημα δεν το απευθύνω σε εσένα, αγαπητέ Σιγητά, το απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε, όπω είπε και εσύ άλλωστε, ότι το Ίντερεκ κυρίω επιτρέπει την συνάντηση μεταξύ των ανθρώπων, τη συνεργασία. Αυτή την παραπάνω ασφάλεια για την Ευρώπη, εγώ δεν την καταλαβαίνω στο προκείμενο πλαίσιο. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή τι είδου περιεχόμενο μπορεί να αποκτήσει. σω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, με διαφωτίσει κάπως περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό το μελλοντικό έργο διαχείριση συνόρων δηλαδή στην ουσία. Είναι λοιπόν θετικό το έγγραφο που έχει καταθέσει και θα συμπληρωθεί με τροπολογίες. Νομίζω ότι μόνο εάν δώσουμε εμείς εδώ ξεκάθαρη και ισχυρή εντολή θα έχουμε και ισχυρή θέση απέναντι στους υπουργού στο Συμβούλιο όταν θα συνεργαστούμε μαζί τους. Σχεδόν τρία λεπτά λέει ο Πρόεδρος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 it is advisable to increase the annual advance payments, which will result in faster reimbursement of beneficiaries' expenses. Further consideration should be given to looking for further amendments simplifying the rules. Thank you. Thank you very much. Mr. Van Miltenburg, you have the floor. Ja, dank u voorzitter. En ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor de hele snelle levering. Want het is niet evident om helemaal in een zomerperiode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 Thank you. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πραγματικά καλή η πρωτοβουλία. Δεν βλέπω την κυρία Άντερσον από την ΚΟΕ. Υπάρχει άλλος ε, εκ μέρους Όχι, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Ροπέ που επίσης δικαιούται τρία λεπτά μια και είναι σκιώδης Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα που πραγματευόμαστε ε, είναι συνειφασμένο και με άλλα θέματα. Εδώ μιλούμε για την περίοδο 2021-2027 και προτείνεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με την κοινωνική συνοχή, τη γεωργία και το καθεξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα με τα κράτη-μέλη, αλλά το ζήτημα που ανακύπτει είναι θα μείνουμε μόνο στα λόγια ή θα περάσουμε επιτέλους και στα έργα. Νομίζω ότι ο συγητής μας μας δίνει μια ξεκάθαρη και πολύ εύστοχη προσέγγιση και είναι προφανές ότι το πρόγραμμα Interreg ήταν πολύ χρήσιμο για όλα τα κράτη-μέλη γιατί το Interreg βοηθά τα κράτη-μέλη να επιλύσουν προβλήματα που δεν μπορούν να τα διορθώσουν με άλλους τρόπους. Είναι λοιπόν ηλίου φαϊνότερο ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση με το παρελθόν. Θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο προπολογισμό του Ίντερεγ. με λυπεί το γεγονός ότι τώρα μιλάμε για τα νέα προβλήματα αλλά δεν προβλέπουμε τα απαραίτητα κονδύλια, νέα κονδύλια και νέους πόρους για να πλήσουμε τα νέα προβλήματα και τις νέες προκλήσεις. Δεν μπορούμε με περιορισμένα μέσα να επιλύουμε όλο και περισσότερες προκλήσεις. Τα κράτη-μέλη και οι εταίροι από τις περιφέρειες ακολουθούν μια χρονοβόρο διαδικασία για να προτείνουν τα προγραμματά τους και είναι συνεχώς σε αγρήγορση, έχουν τις στρατηγικές τους οι διάφορες περιφέρειες και χρειάζεται χρηματοδότηση. Δυστυχώς η χρηματοδότηση όλο και συρρυκνώνεται, κάτι που ε, πλήττει τους πολίτες ε, και τις περιφέρειες που θεωρούν ότι οι επενδύσεις τους δεν έπιασαν τόπο. Θα πρέπει λοιπόν με τα σχόλιά μας να πείσουμε τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο προϋπολογισμό για το Ίντερεκ. Δεν αρκούν τα τρέχοντα κονδύλια. Θα πρέπει να αναζητήσουμε και νέους τρόπους και νέα μέσα χρηματοδότησης. Γιατί μία στρατηγική περικοπής και συρρήκνωσης δεν θα μας βάλει πουθενά. Και θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια διαφύλαξης και ενίσχυσης του Ιντερεκ. Εγώ είμαι της γνώμης ότι το Ιντερεκ είναι απαραίτητο, είναι πολύ χρήσιμο και μάλιστα και προσωπικά είχα ε, μια πολύ θετική εμπειρία με το πρόγραμμα και θεωρώ ότι η εφαρμογή του Ιντερεκ δεν είναι τόσο εύκολη, δεν είναι ε, εξίσου εύκολη με αυτή των άλλων προγραμμάτων. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τους εταίρους μας. Από την άλλη, η διακρατική και η διαπεριφερειακή συνεργασία μας φέρνει πιο κοντά, μας ενώνει και μας επιτρέπει να εμπλουτίσουμε τις εμπειρίες μας. Άρα η προστιθέμενη αξία είναι προφανής. Επίσης, το Interreg προσελκύει επενδύσεις στα διάφορα προγράμματα και επιτρέπει και την ε, ανταλλαγή και αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο λοιπόν το πρόγραμμα και επαναλαμβάνω μας επιτρέπει να λύσουμε πολλά προβλήματα. Όταν εταίροι συναντιόνται συζητούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών επίσης θα είναι πολύ χρήσιμη και καλό θα ήταν να εισακουστεί. Και σε καμία περίπτωση να μην περιοριστεί ο προπολογισμό του Ιντερνετ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω ούτε την κυρία Νταμάτο, ούτε κάποιον άλλο από το κόμμα τη για να μα παρουσιάσει τη θέση του EFTD. Οπότε ολοκληρώσαμε το γύρο με του και οδησηγητές. Δύο άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Η κυρία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 πολύπλοκα τα πράγματα. Δεν βοηθάει καθόλου αυτό σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Υπάρχει το θέμα των, ε, ε, της συνεργασίας με τις θαλάσσιες περιοχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτού του κειμένου. Πολλά από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θαλάσσια και θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Αυτό αφορά το πέμπτο τμήμα στο οποίο η συγητής εκφράζει ορισμένους προβληματισμούς. Πώς θα μπορούσε η Επιτροπή να μας διαφωτίσει, θα μπορούσατε να μας πείτε ένα-δυο πράγματα περισσότερο σε ό,τι αφορά αυτό το τμήμα. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Θα μπορέσει αυτό να γίνει ένα πραγματικό διαπεριφερειακό εργαλείο. Δηλαδή, τι ρεαλιστικές πιθανότητες υπάρχουν να επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις σε συντομία. Το θέμα της ε, προχρηματοδότησης έχει τα Πολύ το δίκιο. Γιατί αν θέλετε να ξεκινήσουμε γρήγορα και αν θέλετε να βοηθήσετε αυτούς ε, τους φορείς, έτσι θα πρέπει να κινηθούμε. Πολλές φορές χρειάζεται το κάψιμο ευθύς εξ αρχής. Υπάρχει λοιπόν ένα λάθος εδώ και θα πρέπει να το διορθώσουμε. Δεύτερον, πραγματικά έχω αμφιβολίες ό,τι αφορά την κριτική σας για το θέμα της καινοτομίας. Γιατί τώρα έχουμε την ε, έρευνα, έχουμε τομεί διάφορους ε, στην έρευνα. Αν διαβάσετε ε, τον ορίζοντα 2020 θα διαπιστώσετε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για Καινοτομία και Τεχνολογία. Ξεκίνησε και αναπτύσσεται ταχαίως. Αυτή η διαπεριφερειακή συνεργασία είναι καθοριστική σημασίας και αν θέλετε να προσεγγίσουν περισσότερο τα ταμεία συνοχής θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την έκτη ταχύτητα. Δεν θα πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι και να αναρωτιόμαστε πώς θα κατανείμουμε τα κονδύλια. Θα πρέπει να επέλθουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογίας. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Νότεμπερκ. Το θέμα είναι το πώς ακολουθούμε τη σωστή τι πορεία προκειμένου να αναπτύξουμε ταχύτητα. Εγώ είμαι συγητήσα ε, για την γνωμοδότηση που αφορά τις συνέργειες μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των κονδυλίων μας. Θα ήθελα να σας κάνω έκκληση, να κινηθούμε προς τα μπρος και όχι να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο, αν όχι θα δώσω το λόγο στο πρόσωπο της Επιτροπής Περιφερειών, που είναι και η συγγήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να πάρω το λόγο και να μιλήσω για το σημαντικό αυτό κανονισμό. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Αριμό, με τον οποίο είχα μία θαυμάσια συνεργασία σχετικά με αυτό το θέμα, ε, ότι ο χρόνος ε, πίεσε πάρα πολύ. Η πρόταση της Επιτροπής συνεπάγεται πολλά θετικά στοιχεία, ιδιαίτερα εμείς στην Επιτροπή Περιφερειών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά τα όσα έχουν γίνει για τις ε, εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή που μίλησε για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την ε, διακρατική συνεργασία για να μπορέσουμε μετά να χρηματοδοτήσουμε τις καινοτομίες στο 5. Επίσης αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει η διατήρηση προγράμματων όπως το ΡΑΤΟ, η ΤΕΡΑΤΑ, θέματα που αφορούν ε, την αναγνώριση της ε, ανάγκης για την υποστήριξη μικρών προγραμμάτων. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε αυτά επί τόπου, γιατί στην ουσία μιλάμε για προγράμματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν επί τόπου. Η Επιτροπή Περιφερειών έχει κάποιο προβληματισμό σε ό,τι αφορά την μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, της τάξης το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπήρξε μία μείωση 42% σε επίπεδο διακρατή κρατική συνεργασίας και η διαπεριφερική συνεργασία έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Μας προβληματίζει επίση επίσης ο διαχωρισμός, όπως ανέφερε ένας συζητητής, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ της διακρατικής συνεργασίας ε, της θαλάσσιας και της χερσαίας. Τα σύνορα είναι σύνορα, είτε ε, σηματοδοτούνται από τη θάλασσα, είτε από ένα βουνό είναι σύνορα και αυτό συνεπάγεται ορισμένα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συνεργαστούν και εκατέρωθε των σύνορων. Ε, επίσης, ό,τι αφορά το Interreg Ευρώπη, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας που βοηθάει τη μεταφορά εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών και θα μπορούσε να επεκταθεί σε περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 174 των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά περιοχές με ιδιαίτερα διαθροτικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, ε, συμφωνώ με τον εισηγητή του Κοινοβουλίου, θα επισημούσαμε μια αύξηση του ποσοστού χρηματοδότης με 80% και η πρόταση όπως διατυπώθηκε να αλλάξει ο υπολογισμός των κονδυλίων του προϋπολογισμού δίνοντας προτεραιότητα στον διακρατικό ε, πληθυσμό ε, σε απόσταση 25 χιλιόμετρων κατά την άποψή μας ε, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά την πτυχή 5 ε, περι, περιφερειακές επενδύσεις, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των ιστορικών πτυχών της συνεργασίας στην Ευρώπη. Με λίγα λόγια, παρόλα που έχει καταγραφεί κάποια πρόοδος, εμείς έχουμε το ίδιο επίπεδο του προπολογισμού, γιατί αυτό συνεπάγεται μια ριζική αλλαγή. Θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση αυτού. Υπάρχει αβεβαιότητα στην Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών πόλεις που εργάζονται, συνεργάζονται στα πλαίσια του Ορμπάκ δεν το καταλαβαίνουν αυτό, δεν το, ε, τα νησιά τα οποία από τη φύση τους έχουν θαλάσσια σύνορα δεν καταλαβαίνουν και εκείνα αυτό νομίζω ότι θα πλήξει την ε, πολιτική εδαφικής συνοχής, ε, τις πρακτικέ συνεργασίας που εδώ και χρόνια έδειξαν την προστιθέμενη αξία της, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Γιατί όλα αυτά τα προγράμματα, όλες αυτές οι δράσεις ε, επέτρεψαν στους ε, λαούς της Ευρώπης να γνωριστούν και πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Για μία ακόμα φορά ευχαριστώ και για την προσοχή σας και την προσκλησή σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Μοπερτή. Μας παρουσιάσατε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κιγιώμη, για να μα παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να απαντήσει τις ερωτήσεις ε, που υπευλήθησαν και ίσως μας δώσει και κάποιες εξηγήσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης του και τους ε, ευρωβουλευτές που σχολίασαν την πρόταση, καθώς και την εισηγητήρια της Επιτροπής των Περιφερειών, την κυρία Μαπερτουή. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το Interreg και την ε, θερμή υποστήριξη που το επιφυλάξατε. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των ε, ομιλητών ε, τάχθηκαν υπέρ του Interreg. Και επίσης χαίρομαι που υποδεχθήκατε θερμά τα νέα στοιχεία που υποβάλαμε για το Interreg. Τώρα για τα γενικά χρηματοδοτικά κονδύλια για το ΙΝΤΕΡΕΚ θα πρέπει να τα δούμε στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στο συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο μετά το 2020. Δεν θα σταθώ λοιπόν στα γενικά στοιχεία, αλλά θα επισημάνω μια αντίφαση που ακούσαμε. Γιατί από τη μια ζητάτε αύξηση του προπολογισμού του Ιντερεκ, που δεν συμβιβάζεται με την πρόταση ε, της τροποποίησης ε, του συντελεστή συγχρηματοδότηση από το 70% στο 85% γιατί έτσι θα μειωθεί γενικώ το ποσοστό διαθέσιμων επενδύσεων για το ΙΤΕΡΑ και ο κύριος Μίλτεμπορκ ε, πολύ σωστά το επισήμανε. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό γιατί ε, πολύ σωστά και εύστοχα τα παρουσίασε ο κύριος Μίλτεμπερκ με τον οποίο συμφωνούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια συνεργασία, που φαίνεται ότι προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε ούτε περικοπή ούτε διακοπή της στήριξης στην θαλάσσια συνεργασία. Προτείνουμε απλώς αλλαγή της μεθόδου λειτουργίας της θαλάσσιας συνεργασίας. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αναγνώριση που κάνουμε της ε, διαφορετικής φύσης που έχει η θαλάσσια συνεργασία σε σχέση με τη χερσαία συνεργασία. Όπως επισήμανε και οι πρόσωπο τη Επιτροπή των Περιφερειών, το σύνορο είναι σύνορο, είτε είναι χερσαίο είτε είναι θαλάσσιο. Άλλο όμω τα χερσαία σύνορα και άλλο τα θαλάσσια σύνορα, ω προ το είδο τη συνεργασία που θα μπορούσαμε να στηρίξουμε και του τομεί ε, ε, συνεργασία, του οποίου θα μπορούσαμε να δώσουμε προτεραιότητα στην α ή β μορφή συνεργασίας, αν έχει χερσαία δηλαδή θαλάσσια. Επίσης θέλουμε ένα πιο ολοκληρωμένο και συντονισμένο πακέτο συνεργασίας, ιδιαίτερα στις ε, θαλάσσιες λεκάνες, συνδυάζοντας ε, την μέχρι στιγμής παραδοσιακή διμερή θαλάσσια συνεργασία και συνδυάζοντας την πιο αποτελεσματικά με την συνεργασία στις μακροπεριφέρειες ή στις θαλάσσιες λεκάνες. Γι' αυτό και υιοθετούμε διαφορετική προσέγγιση για να θετήσουμε μια πιο στρατηγική και πιο ευρεία προσέγγιση. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είχε μόνο υπέρμαχος μια τέτοια αλλαγή της προσέγγιση, αλλά πιστεύω ότι έτσι θα ενισχύσουμε τη συνεργασία και θα προ... σημειώσουμε πρόοδο στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Επίσης, για, τις... για το σημείο 5, σε 5 των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία. Ε, σημειώνουμε τα σχόλιά σας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η συνιστόσα εντάσσεται πολύ αρμονικά στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του Ιντερεκ, ακριβώς γιατί εστιάζεται στην διαπεριφερειακή συνεργασία και αξιοποιεί το βασικό στοιχείο της ε, πολιτικής συνοχής των τελευταίων χωρών, δηλαδή την ε, ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση στρατηγικών ε, ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και δίνοντας έμφαση στις αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών. Πολύ επίσης επισήμανα την ανάγκη πολιτική καινοτομία γενικώ, αλλά και η πολιτική καινοτομία της ε, συνοχής να είναι πιο εξωστρεφής και να επιδιώκει καλύτερες Καλύτερου δεσμού μεταξύ των περιφερειών. Επίση θέλουμε να αναπτύξουμε αλυσίδε αξιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και να ενισχύσουμε του δεσμού και τη συνεργασία του με άλλε περιφέρειες στι πιο ανεπτυγμένε περιοχέ τη Ευρώπη. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χάρη σε στοχευμένε δράσει, που ε, θα ε, υποβοηθούνται μέσω ε, της άμεσης διαχείρισης και όχι της προσέγγισης των προγραμμάτων στις ε, καινοτόμες δράσεις του Urban τέτοιου είδους ε, εστίαση. Έχουμε στη διακυβέρνηση και επίσης να επικεντρωθούμε περισσότερο στη μέθοδο αποτελεσμάτων παρά ε, στις επιδιώξεις μας και τους στόχους μας. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για τη διάσταση της ασφάλειας που επισημάνατε. Αυτό συνδυάζεται και με την συμπερίληψη της συνιστώσας του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων που μπήκε ε, πια ρητά στον κανονισμό. Και αυτή είναι προτεραιότητα και στα εφιστάμενα προγράμματα ε, των, ε, της διαχείρισης εξωτερικών συνόρων που εμπίπτουν σε διάφορους κανονισμούς σήμερα. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί η διάστηση της ασφάλειας εκεί που χρειάζεται σε κάποια εξωτερικά σύνορα. Οπότε προσφέρεται ως μη επιπλέον ε, δυνατότητα για παροχή βοήθειας και υποστήριξης. Και θα τελειώσω με δύο ίσονο σημασία ζητήματα. Καταρχήν τα ποσοστά σφάλματος και το πώς επηρεάζουν το ίντερεκ. Ένας από τους λόγους για την αλλαγή της προσέγγισης που προτείναμε για τους ελέγχους σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Interreg είναι γιατί όταν ε, εξετάζουμε το συνολικό αντίκτυπο του Interreg, διαπιστώνουμε ότι έχει σταθερά χαμηλά ποσοστά σφάλματος. Αν ε, δούμε το Interreg ως πακέτο προγραμμάτων, υπάρχουν κάποιες επιμέρους δυσκολίες σε μεμονωμένα προγράμματα, αλλά αν δούμε το Interreg ως σύνολο, το υψηλότερο ποσοστό σφάλματος που έχει καταγραφεί σε συγκεκριμένη χρονιά είναι 1,6%. Οπότε είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι γενικά τα προγράμματα του Interreg δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με σφάλματα, με ποσοστά σφάλματος. Και γι' αυτό προτείναμε να ομοδοποιήσουμε τα προγράμματα και να τα α, αντιμετωπίσουμε ως ενίο πακέτο. Έτσι θα μειωθεί αισθητά το, το βάρος του ελέγχου σε όλα τα, τα προγράμματα. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θα ήθελα να το ξεχωρίσω. Το επισήμανε και η κυρία Μοπερτουή. Αφορά τη νέα συνιστόση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Εκεί φροντίσαμε να έχουμε κατάλληλο προϋπολογισμό για τα προγράμματα των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να συνεχίσουν το έργο τους και να συνεχίσουν την πορεία τους προς την πρόοδο. Και μάλιστα η πρόταση του, του του μειώνει τον προπολογισμό αυτό σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδα και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί και δεν είμαι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο θα το περιμέναμε από την Επιτροπή σας. την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μας ευνηδίασε Μάλλον αρνητικά και θα ήθελα να το έχετε υπόψη για τι μελλοντικέ συζητήσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα ο λόγο στον εισηγητή, του κ. Ρημό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Τα σημείωσα όλα όσα άκουσα και θα τα περιλάβω κατάλληλα στο κείμενό μου. Αναμένω με ενδιαφέρον τι τροπολογίε που θα καταθέσουν οι συναδελφοί μου. Ένα θέμα που θέλω να σχολιάσω σύντομα είναι αυτή η συνιστόσα 5, component 5. Εάν εκπροσωπούμε την άποψη, όπως νομίζω όλοι εκπροσωπούμε, ότι δεν θέλουμε να ρεύσουν λιγότερα κονδύλια στο Ιντερεγ, λιγότερα από όσα μέχρι τώρα, γιατί θέλουμε να λειτουργήσουν τα προγράμματα Ιντερεγ το ίδιο καλά όπως έως τώρα. Δεν θα πρέπει λοιπόν τότε να δεχθούμε είτε να πούμε ίδιοι ότι συμφωνούμε ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τα κλασικά αυτά προγράμματα να περικοπεί. Διότι αυτό σημαίνει να δεχθούμε την συνιστόσα 5. Εγώ δεν είμαι αντίθετο με τη συνιστόσα 5 και με τα όσα προτίθεται να χρηματοδοτήσει. Συμφωνώ να γίνουν. Αλλά πρέπει αυτό να γίνει σε βάρο των άλλων προγραμμάτων που έω τώρα έχουν λειτουργήσει καλά. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτω. Εγώ θα έλεγα μακάρι να δοθούν 5 δισεκατομμύρια στην σε αυτή αν η Ευρώπη πράγματι θέλει να γίνει πρωτοπόρος σε κάποιες τεχνολογίες. Αλλά να γίνει αυτό εις βάρος του προϋπολογισμού Interreg, αυτό σημαίνει ότι στην ουσία τιμωρούμε εκείνους οι οποίοι μέχρι τώρα έδρασαν και λειτουργήσαν με επιτυχία η προηγούμενη περίοδος είχε φτάσει 9,3 δισεκατομμύρια. Τώρα είμαστε στα 8,4. Αν αφαιρέσουμε άλλο ένα δισεκατομμύριο από αυτά τα 8,4 και τα βάλουμε στην component 5, τότε βρισκόμαστε στα 7,4. Δηλαδή μείωση τελικώς κατά 21%. Άμα θέλετε να βγείτε να το πλασάρετε αυτό έξω, τι να σας πω, καλή τύχη. Εγώ είμαι υπέρ του Interreg, θέλω να παραμείνουν τα προγράμματα αυτά, να διατηρηθούν, διότι πρόκειται για θετικό μήνυμα υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας πολύ ευχαρίστω να διατηρηθεί η συνιστόσα 5, αλλά να δοθούν νέα, να ενωθεί νοπό χρήμα για αυτήν. Εγώ προτείνω 0,3% για την ε, συνιστόσα 5. Αυτά όμως πρέπει να προέλθουν από τις χώρες μέλη τα χρήματα αυτά. Όχι σε βάρος των παλαιών κλασικών προγραμμάτων Interreg. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάθεση τροπολογιών. Μιλήσατε πριν, κυρία Πρόεδρε, για τις 17 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίρρηση από κανένα. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλες και όλους για τα σχόλια και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την περαιτέρω συνεργασία. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύντομος χρόνος δηλαδή, πολύ σύντομος. Αν μπορεί να δεχθεί λοιπόν και ο εισηγητή να αναβάλουμε την προθεσμία αυτή για τι 17 Ενάτου, 17 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα λοιπόν, το δέχεστε, ωραία. 17 Σεπτεμβρίου προθεσμία υποβολή τροπολογιών για τη σημαντική αυτή έκθεση του κυρίου Αριμών. Σα ευχαριστώ πολύ για την γόνιμη συζήτηση, ευχαριστώ και του προσκεκλημένου. Σα εύχομαι καλή επιτυχία στην εργασία σα που δεν θα είναι εύκολη κύριε Αριμών. Τώρα να ευχαριστήσω την κυρία Μπρέσο, η οποία μετακινείται μεταξύ επιτροπών και βλέπω ότι ήρθατε ακριβώς την ώρα για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την συζήτηση για τη γνωμοδότησή μας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι ο βασικός μηχανισμός της Ευρώπης για την στήριξη των ανθρώπων για να βρουν καλύτερη δουλειά, να βρουν δουλειά, να βρουν καλύτερη δουλειά, να δοθούν ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Από τις 29 Πέμπτου φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το νέο κοινωνικό ταμείο Plus. Η Επιτροπή Απασχολήσεω είναι καταρχήν αρμοδία επί για το ταμείο αυτό. Η δική μας ωστόσο Επιτροπή έχει ορίσει ω εισηγήτρια την κυρία Μπρέσο για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεω. Σήμερα η κυρία Μπρέσο θα αναπτύξει το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδοτήσεώς της και για αυτό το λόγο της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή μιλάμε για νομοθετικό κείμενο, θα ήθελα να παρουσιάσω μια σύντομη αιτιολογική έκθεση και μια σειρά τροπολογιών που αφορούν το κείμενο και που θα πρέπει να διαβιβαστούν στην αρμόδια επιτροπή. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή στην πρόταση που αφορά το νέο κοινωνικό ταμείο, το οποίο ονομάζεται FSA SIN Plus, ενώνει όχι μόνο το παραδοσιακό κοινωνικό ταμείο, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το, ε, το, τα προγράμματα για κοινωνικές ε, Καινοτομίε και το πρόγραμμα WAVE ε, για την υγεία. Και βεβαίως αυτό ανήκει τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει ο περιφερειακός χαρακτήρας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ότι στην αρμόδια επιτροπή υπάρχουν ορισμένοι προβληματισμοί σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος για την υγεία, που φαίνεται να μην συνάδει τόσο πολύ με το υπόλοιπο ταμείο, με τους στόχους του κοινωνικού ταμείου. Βεβαίως, εκφράζουμε τη σύμφωνη γνώμη μας στην γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά το ρόλο του κλειδί που θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει το κοινωνικό ταμείο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, κατάρτισης, προώθησης της κοινωνικής ένταξης αλλά και θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτή τη διεύρυνση σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης. Εκεί υπάρχει ένα ποσοστό 25% και ένα 2% για την καταπολέμηση της ε, έλλειψης υλικών αγαθών. Εδώ μιλάμε για άτομα τα οποία ούτε καταρτίζονται, ούτε εργάζονται, ούτε σπουδάζουν και στα άτομα αυτά δίνεται το, το 10% θα πρέπει να δίνεται σε πολιτικές για απασχόληση νέων. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά αυτό το σημείο. Βεβαίω δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, οι ενεργείες πολιτικές για την ένταξη στην ομάδα εργασίας παραμένουν ο πυρήνας του κοινωνικού ταμείου και θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι. Ένα πρώτο σημείο που μας αφορά ως Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων είναι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται ρητά στο κείμενο ο ρόλος των περιφερειών και αυτό θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος γιατί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών για την απασχόληση και την κατάρτιση και των εργοπολιτικών πολιτικών εργασίας από τη μία και των πολιτικών ανάπτυξης που προωθούνται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να συνεχίσουν να υφίσταται γιατί στην ουσία είναι οι, ίδιο, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μία σειρά από τροπολογίες καθιστούν σαφές ότι δεν μπορεί να πάψει να υφίσταται αυτή η σχέση, δεν μπορεί να εθνικοποιηθεί το SSA πλάσα και να παραμείνει η περιφερειοποίηση του τέταρτου. Δηλαδή και τα δύο τα ε, ταμεία τα πρέπει να συνεχίσουν να ανήκουν στον ίδιο προγραμματισμό όπως έχει γίνει για από τις περιφέρειες. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η παρατήρηση έγινε και στην Επιτροπή ΕΜΠΛΕ. Και οι τροπολογίες μας θα μπορούσαν να τύχουν θετικής υποδοχής. Υπάρχουν μία σειρά από απλουστεύσεις που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε θα έλεγα. Γιατί πιστεύουμε ότι καθίσταται περισσότερο εφικτή πραγματοποίηση η επίτευξη των στόχων. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας όχι μόνο στα θέματα που αφορούν το ρόλο των εθνικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων, θεσμών, με συγχωρείτε, ε, αλλά τη συνοχή μεταξύ όλων των διαρθρωτικών ταμείων. Δηλαδή όλα τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει, και όλα τα άλλα εργαλεία θα πρέπει να ανήκουν σε ένα και μοναδικό πακέτο που θα αποτελεί αντικείμενο ενός σωστού σχεδιασμού. Το δεύτερο σημείο, κατά την άποψή μου, σημαντικό σημείο, ένα σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει μέσω των κανονισμών, αφορά την συνοχή μεταξύ του νέου πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όχι μόνο τους παραδοσιακούς στόχους των πολιτικών συνοχής, αλλά και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τα προβλεπόμενα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για τις μεμονωμένες χώρες. Το θέμα είναι ότι ο συνυπολογισμός των πολιτικών αυτών συνδέεται άμεσα με τον πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό, το, η Προεδρία θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει υπόψη της και τις κοινωνικές πολιτικές και την ανάγκη για βελτίωση αυτών των πολιτικών στα πλαίσια των προβλεπόμενων για την κάθε χώρα όπως έχουμε τονίσει και σε άλλα κείμενα. Δηλαδή αυτές είναι οι πτυχές του συγκεκριμένου εξαμήνου ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κοινωνικό ταμείο. Ο, ε, το εξάμεινο αυτό το εξάμεινο αυτό γίνεται προγραμματισμός ετήσιος. Εμείς μιλάμε για ε, προγραμματισμό 7 ετών. Αναφέρεται εδώ ότι η συνοχή θα πρέπει να επιτυχάνεται μόνο στην αρχή της περίοδου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και στο ίμιση της εντολής το ίμιση της περίοδου προγραμματισμού όταν γίνεται η αναθεώρηση. Όχι κάθε χρόνο, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε μια ριζική αλλαγή της ε, δομής των διαθροτικών ταμείων και συγκεκριμένη περίπτωση του κοινωνικού ταμείου. Βεβαίως, θα πρέπει όλα αυτά που προβλέπουμε να ε, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους στόχους. Δηλαδή το στοιχείο της ολοκλήρωσης να υπάρχει στο ευρωπαϊκό εξάμεινο σε ό,τι αφορά τους στόχους που συλλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό ε, πυλώνα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτό αφορά μόνο την Ιταλική μετάφραση Στην τροπολογία 1, ε, στην ε, αγγλική μετάφραση, για λόγους που δεν κατάλαβα, έχουν συμπτυχθεί δύο τροπολογίες. Η σωστή μετάφραση είναι η αγγλική. Τροπολογία 12 σε άλλες γλώσσες παρατίθεται ως τροπολογία 11. Τώρα φαντάζομαι ότι θα διορθωθεί μετάφραση στα Ιταλικά, γιατί όπως σας είπα δεν έχει σχέση με αυτό που έγραψα στα Αγγλικά, γιατί το κείμενο ψηφίστηκε στα Αγγλικά. Δεν ξέρω πώς είναι στις άλλες γλώσσες. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να διορθώσουν την τρομπολογία 12. Δηλαδή αν θέλουν να, κάνουν, ε, να υποβάλουν κάποια τροπολογία να αναφερθούν στο αγγλικό κείμενο. Αυτό αφορά, αφορά το περιεχόμενο της τροπολογίας. Ε, συγγνώμη που παρεξέκλεινα, αλλά ε, ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ των αγγλικών και των ιταλικών. Εγώ ήθελα απλώς να σας το πω, ρίξτε ματιά στα αγγλικά για να το δείτε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπρέσο. Φαντάζομαι θα διευκρινιστεί αυτό το ένιγμα μεταξύ των τροπολογιών 11, 12 και 18. Όχι, 11 και 12. Το 12 στην αγγλική μετάφραση είναι η τροπολογία 11 στην ιταλική. Και δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η αναντιστοιχία. Καλά, θα το φροντίσει η γραμματεία να εφηγραμμιστούν οι αριθμίσει των τροπολογιών σε όλε τι μεταφράσει. Ευχαριστώ και περνάμε στου κοιόδη ηγητέ και να δώσω πρώτα το λόγο και μετά φυσικά στα μέλη τη Επιτροπής ΡΕΚΙ και σα θέλω παρακαλώ και πάλι να τηρήσετε το χρόνο σα. Τρία λεπτά έχει ο κάθε σκιώδης ηγητή και θα δούμε μετά για του υπόλοιπου. Ο κύριος Χέτμαν απουσιάζει. Ποιο θα τον αντικαταστήσει, ο κύριο Όλμπριχτ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα διαβάσω στα πολωνικά τα σχόλια του κυρίου Χέτμαν, γιατί καθυστέρησε η πτήση του, βρίσκεται ακόμη στο αεροπλάνο ο κύριο Χέτμαν. Θα διαβάσω λοιπόν στα πολωνικά. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστώ την κυρία Μπρέσο, τη εισηγητρία, για την ισορροπημένη και αξιόλογη γνωμοδότησή της. Συμφωνώ με τις βασικές προτάσεις και προσεγγίσεις της για το νέο ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συμφωνώ με την καλύτερη διευκρίνηση του ρόλου των περιφερειών και την υπογράμμιση τους, γιατί όχι μόνο είναι δικαιούχοι οι αλλά και διαχειριστικές αρχές ε, του ενισχυμένου ΕΚΤ, αλλά έχουν και περισσότερες ε, γνώσεις και πολύ χρονή πείρα για τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πολύ σωστά λοιπόν και εύστοχα το επισήμανα η συγγετρία, γιατί σίγουρα ο του περιφερειού θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του ενισχυμένου ΕΚΤ. Με ικανοποιεί και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση της εφαρμογής του ενισχυμένου ΕΚΤ, του ΕΚΤ-ΣΥΝ. Επίση, ε, ή ο συνδυασμός των διαφόρων μέσων θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης του ενισχυμένου ΕΚΤ. Ε, θα πρέπει όμως για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος ε, να έχουμε κοινέ ε, διατάξεις για την εφαρμογή των διαφόρων μέσων. Επίσης καλό θα ήταν να συμβάλλουμε ώστε οι ειδικοί στόχοι να εξυπηρετούν και τους γενικούς στόχους και να επικεντρωθούμε στα βασικά θέματα της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης. Θεωρώ όμως ότι το ΕΚΤΣΥΝ θα πρέπει να δώσει περισσότερη σημασία στα δημογραφικά προβλήματα και σε εδαφικό πλαίσιο, γιατί οι εξόχως απόκεντες περιοχές είναι οι πιο αεροκατοικημένες και παρουσιάζουν περίμωση και να λάβουμε υπόψη και το θέμα της γύρασης του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Επίσης, ε, ε, με στενότερη συνεργασία του ΕΚΤ με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, θα βελτιώσουμε την καλύτερη δρομολόγηση και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Βέβαια, θα πρέπει να διευκρινίσουμε πολλά άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ε, ποια συγκεκριμένα προγράμματα θα, θα ε, προωθηθούν από τα κράτη-μέλη και τι γίνεται σχέση με τα λειτουργικά προγράμματα. Θα πρέπει να ε, έχουμε καλύτερο συντονισμό του πολυετούς ε, κύκλου λειτουργίας του ΕΡΚ και των μονοετών κύκλων συγκεκριμένων προγραμμάτων. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολύ λογική και ισορροπημένη η πρόταση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και η, γνώση της, και η πρόταση της εισηγήτριας και έχουμε μια πολύ καλή βάση για εργασίας. Πιστεύω ότι θα είναι αποτελεσματικές οι εργασίες μας και θα καταλήξουν σε μια αξιόλογη γνωμοδότηση τη Επιτροπή ΡΕΚΙ προς την Επιτροπή Απασχόλησης που είναι η καθήλη αρμόδια. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φίτο απουσιάζει όμω τον αντικαθιστά κυρία Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ. Το ECR αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ε, έξυπνη εξειδίκευση, τη διαβίου κατάρτιση και τα μοντέλα κατάρτιση με δικαιούχου κυρίως του νέους που βρίσκονται εκτός απασχόληση εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και τους εκπαιδευτέ, ε, εκπαιδευτικού, προπονητέ, ερευνητέ ε, και επιχειρηματίε θεωρούμε ότι ο σαφή ρόλο των περιφερειών και ω δικαιούχων και ω διαχειριστικών αρχών θα πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα στο νομοθετικό κείμενο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των στόχων που αναφέρονται στην πρόταση και να εξασφαλιστεί ε, κατάλληλο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΤΣΥΝ της εδαφικής συνοχής, ε, της περιφερειακής πολιτικής και των χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης, χαιρετίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλουστεύσει το νομοθετικό πλαίσιο και θεωρούμε ότι οι συνέργειες και ο συντονισμός μεταξύ του ΕΚΤΣΙΝ και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αύξησης της αποδοτικότητας στην υλοποίηση των στόχων του ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαμίλτεμπορκ είναι ο επόμενος και ηγετής. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Μπρέσο για την ταχύτητα με την οποία διεκπαιρέωσε το έργο της και την πολύ αξιόλογη γνωμοδότησή της. Συμφωνώ, 10% των κονδυλίων να δοθούν ε, για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ποσοστό θα πρέπει ε, οι νέοι είτε να εργάζονται, είτε να σπουδάζουν, είτε να, κάνουν κάποια, να παρακολουθούν κάποια σεμινάρια, ε, κάποια κατάρτιση. Γι' αυτό είμαι υπέρ του ποσοστού του 10% για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όπως είπα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχασε μια σημαντική ευκαιρία να ενισχύσει ε, την συνοχή με τη συμπερίληψη και τη συγχώνευση στο ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κρίμα που δεν έγινε η συγχώνευση και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στο νέο ΕΚΤ. Ε, κρίμα γιατί από τη μια ζητάτε απλούστευση και από την άλλη την αποφεύγετε ναι, μεν περιλάβατε το πρόγραμμα για την υγεία ή το πρόγραμμα προς τους απόρους ή την κοινωνική καινοτομία. Τι γίνεται όμως με μια επιχείρηση που για τον α ή β λόγο θα χρειαστεί να κάνει μαζικές απολύσεις σε χώρες που υπάρχουν, σε περιοχές που υπάρχει υψηλή ανεργία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε προγράμματα απασχόλησης ή κατάρτισης ή προγράμματα καινοτομίας. Η καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Χάρη στην καινοτομία θα μπορέσουν πολλοί συνάνθρωποι μας να ξαναβρούν μια θέση εργασίας. δεν θα πρέπει να συνεχίζουμε να βάζουμε γύψο σε ένα ξύλινο μέλο. γιατί αυτό το ρόλο κάνει τελικά το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Κρίμα που δεν συγχωνεύτηκε με το ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χάσατε μια πολύ σημαντική ευκαιρία, θα ήθελα να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, το συνολικό κονδύλιο μειώθηκε, ενώ απ' την άλλη βρισκόμαστε μέσω μια δημογραφική κρίση και μια γύραση του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα κονδύλια στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχες συνέργειες ε, με το νέο πρόγραμμα για ορίζοντας Ευρώπη, κάτι που δεν ε, το βλέπω στην τελευταία πρόταση. Και το 2% των εθνικών κονδυλίων που υποτίθεται θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ε, εξαθλίωσης αρκεί αυτό το ποσοστό, μόνο 2% και θα πρέπει να περάσουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο για να το επιτύχουμε. Δεν είναι καλύτερο να αφήσουμε αυτό το ζήτημα στα κράτη-μέλη, γιατί η εξάλληψη της φτώχειας θα πρέπει να γίνει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, κοντά δηλαδή σε αυτούς που βρίσκονται στο όριο της εξαθλίωσης και της φτώχειας. Σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της ένδυας και της εξαθλίωσης δεν ενθουσιάστηκα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να με συμβολικά να έχουμε μια θετική πρόταση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και εμπράκτος και αν όντως θα οδηγήσει σε καταπολέμηση της φτώχειας ίσως θα πρέπει να ενισχύσουμε κάπως την γνωμοδότηση. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι είναι θετική η προσέγγιση της και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε μια καλή γνωμοδότηση στην Επιτροπή Απασχόλησης και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους και εισηγητές. Η κυρία Νταμάτο απουσιάζει. Άλλος κανείς από το EFTD? Όχι. Άλλα σχόλια υπάρχουν. Ο κύριος Βανίστερόι. Ευχαριστώ πολύ. Στην πρώτη συνάντηση καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Και με λυπεί το γεγονό ότι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό σε επενδυτικοποίηση. Υπάρχει ο κοινωνικός πυλώνας και αυτό είναι το τέλος των ε, εθνικών κρατών. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία έχουμε το περιφερειακό ταμείο και υπάρχει και η επιρροή των πόλεων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα εθνικό πρόγραμμα. Αν λέτε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί Εάν δεν κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα. Εσείς αναφερθήκατε στις γενικές πολιτικές. Ε, θα ήθελα να πω ότι τα επτά χρόνια θα πρέπει να μας απασχολήσει ο πληθυσμός ο Ρωμά. Θα πρέπει, έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα. Αν δούμε πόσα χρήματα έχουν επενδυθεί, θα καταλάβουμε ότι δεν επιτύχαμε το στόχο μας. Δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει μετανάστευση. Θα πρέπει να υπάρχουν, ε, να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, πραγματικά καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αποδοτικοί. Θα πρέπει να, δοθούν, να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια στο κοινωνικό ταμείο και σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θυμάμαι ότι την περίοδο αυτή είπαμε ότι θα υπάρχουν χρήματα που θα εισρεύσουν σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να δοθούν και καλύτερα σημεία για να ε, οικοδομηθούν καινούργια σπίτια. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό στην έκθεση Μπρέσο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στη γυρία σου κουβατός εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους ε, εισηγητές και όδες εισηγητές. Πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που και θα τις λάβουμε υπόψη μας. Θέσατε το θέμα του πρωταετούς προγραμματισμού και του κοινωνικού πυλώνα. Αυτό πλύνεται από την πρόταση για προγραμματισμό του 5 συν 2. Αυτό επιτρέπει μία ενδιάμεση αναθεώρηση κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά το ίδιο το εξάμεινο θα είναι ένα άτυπο εξάμεινο. Ε, το 2020 και το 2019 οι συστάσεις των χωρών χρησιμοποιούνται και εκθέσεις χρησιμοποιούνται ως βάση για προτάσεις στα κράτη-μέλη προκειμένου να δουν πού θα πρέπει να γίνουν αυτές οι προτάσεις για επενδύσεις. Θα υπάρχουν δύο εξάμεινα από ό,τι γνωρίζουμε τώρα Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνο εθνικοποίηση των πολιτικών, γιατί οι κανόνε για εφαρμογή βρίσκονται στον κοινό κανονισμό, αφήνουν περιθώριο για περιφερειακά προγράμματα και εξασφαλίζουν τη συνέχιση ε, ώστε να υπάρχει ένα ε, ε, ε, διαφορετικό επίπεδο προγραμματισμού. Νομίζω ότι οι διαχειριστικές αρχές θα μπορούσαν σε διαφορετικό επίπεδο, αλλά εδώ μιλάμε για οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα για την Επιτροπή, ότι υπάρχει μια διαχειριστική αρχή σε πολλά επίπεδα. Πιστεύω ε, ε, βεβαίως αναμονήσαμε τους κανόνες για εφαρμογή. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δημογραφικές αλλαγές, στις ε, περιοχές ε, οι οποίες είναι εξόχως απόκεντρες θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ίδιες δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές από τις παρεμβάσεις είναι πιο ακριβές λόγω της απόστασης. Δεν έχουμε να κάνουμε μια καινούρια σειρά μέτρων. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παραδοσιακά μέτρα για να μπορέσει να γίνει η άμεση εφαρμογή. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει ένα προληπτικό εργαλείο προκειμένου να μπορεί έγκαιρα να αντιμετωπίζει προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοηθάει τους ανθρώπους που ήδη απασχολούνται να αποκτήσουν νέα προσόντα, νέες γνώσεις, έτσι ώστε να μην απολυθούν. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αφορά μία εκ των υστέρων παρέμβαση. Υποστηρίξουμε άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους με συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένη στήριξη και η πρόταση της Επιτροπής είναι να διατηρηθεί αυτό το εργαλείο και να δοθούν επιπλέον δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αντιδράσουν άμεσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να υποστηρίξει εταιρείες όταν χρειάζεται αναδιάρθρωση, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης έχει άμεση συμμετοχή στην παροχή βοήθεια προς τους ανθρώπους. Σε ό,τι αφορά το θέμα του προγράμματος ε, υγείας, Μπορώ να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας είναι ένα εργαλείο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε, να υιοθετήσουμε μια πειραματική προσέγγιση που να αφορά όλες τις χώρες μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που αλλάξουν το σύστημα υγείας. Και ε, το ποσό είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί παράδειγμα και σημείο αναφοράς και όταν αυτά τα καλά αποτελέσματα ή τα ε, ε, καλά προγράμματα εφαρμοστούν στις χώρες μέλη θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για νέες συνέργειες αλλά και για το ίδιο το Κοινωνικό Ταμείο σε ό,τι αφορά το θέμα των Ρωμά δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Γι' αυτό μιλήσαμε για ένταξη όχι 20 αλλά 25%. Ε, το θέμα μας δεν είναι μόνο η ενσωμάτωση των Ρωμά. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Πιστεύουμε ότι το 25% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να αφορά την ε, ε, ένταξη των Ρωμά. Το, ε, θα πρέπει να συνεχίσει να παράγεται στήριξη σε ανθρώπους ε, που έχουν πολλές ανάγκες, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να διανύσουν μια δύσκολη περίοδο και να μπορούν να, να τρέψουν στα μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορούν τα μέτρα αυτά ένταξη στην αγορά και ένταξη στην κοινωνία θα πρέπει να δοθούν, να δοθεί ηλική υποστήριξη στους ανθρώπους και μετά να τους προσφέρουμε περισσότερο απτή υποστήριξη για το μέλλον. Ευχαριστώ. Α, ευχαριστώ παρακαλώ. Η κυρία Μπρέσο αν θέλει να επανέλθει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους Νομίζω ότι θα μπορούσα να πω ανακεφαλαιώνοντας ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της μεγαλύτερης σύνδεσης με τις περιφερειακές πολιτικές, δηλαδή το θέμα ότι τουλάχιστον το σημαντικό, για το σημαντικό κομμάτι του Ταμείου θα πρέπει να διατηρηθεί σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συμφωνούμε. Αν κατάλαβα καλά, η Επιτροπή συμφωνεί λίγο λιγότερο το να αφήσουμε ελεύθερα τα κράτη να αποφασίσουν είναι κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνη γιατί μπορεί να υπάρχει μία βασική αποσύνδεση μεταξύ δύο ταμείων. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεργάζονται τα δύο αυτά ταμεία. Δεύτερο, οι παρατηρήσεις που διατύπωσε ο συνάδελφος Μούλτεμπεργκ Καταλαβαίνω ότι είναι σωστό να λαμβάνει υπόψη στη χρήση ε, του Ταμείου ε, του Περιφερειακού Ταμείου και του Κοινωνικού Ταμείου, είναι σωστό λοιπόν να, να λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη προσαρμογής της επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Όπως όμως αναφέρθηκε, αυτό είναι ένα ταμείο που διαχειρίζεται η Επιτροπή εκτός του πολιετούς προγράμματος ενδεχομένως ε, ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια υπόμνηση της ανάγκης συντονισμού. Μπορούμε όμως να το βάλουμε εδώ. Με χαρά λαμβάνω υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις συγκεκριμένες συστάσεις. Μόνο τα δύο αυτά χρόνια, το χρόνο εκκίνησης και το χρόνο αναθεώρησης, θα, ληφθούν, θα ληφθεί η υπόψη τη μία, στιγμή αυτή προγραμματισμού του ε, Ταμείου, ε, ε, ε, του Ταμείου. Εμείς ε, θα το κάνουμε, αλλά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη μετέπειτα εξέλιξη του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, γιατί αυτό εδώ συμπεριλαμβάνει και θέματα κοινωνικά, αλλά στο δικό του πλαίσιο, έτσι ώστε να υπάρχει, υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν το κοινωνικό ταμείο στις ε, συστάσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων, εμείς θα συνεργαστούμε προκειμένου να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Και το τελευταίο μήνυμα σε αυτή τη συζήτηση είναι η διορία για τις τροπολογίες που λύγει στις 14 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. 14 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, λίγη διορία για την υποβολή τροπολογιών. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. 14 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την γνωμοδότηση της κυρίας Μπρέσο. Και περνάμε στο επόμενο θέμα. Γνωμοδότηση επίσης την θέσπιση του μηχανισμού ή της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη που προωθεί την απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και επενδύσεις στις μεταφορές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες και στις σχετικές υποδομές. Στην πρόταση αυτή για την επόμενη γενιά του συνδέοντος στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει παράταση του προγράμματος με επιπλέον κονδύλια και ευρύτερο πεδίο εφαρμογή. Η Ήτρε και η ΤΡΑΝ είναι οι συναρμόδιες επιτροπές δυνάμει του άρθρου 55 και θα συντάξουν μια πολύ σημαντική έκθεση, ενώ η δική μας επιτροπή θα συντάξει γνωμοδότηση για την οποία διόρισε τον κύριο Πιοτρόφσκι από το ECR για να την συντάξει. Σήμερα θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση του συντάκτης της, ο κύριος Πιοτρόφσκι που όμως δεν έχει έρθει ακόμη, θα πρέπει να τον περιμένουμε λίγο, αλλά θα καταφτάσει ένα πάσα στιγμή. Βρίσκεται σε άλλη επιτροπή μάλλον. Λίγα λεπτά λοιπόν υπομονή, μέχρι ότου έρθει ο συντάκτη τη γνωμοδότησής μας. Να σας υπενθυμίσω την προθεσμία για τις τροπολογίες που λέγει το μεσημέρι της παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Λιγότερο από μια εβδομάδα λοιπόν έχετε για να υποβάλλετε τροπολογίες για την γνωμοδότηση είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να ε, σεβαστούμε και το χρονοδιάγραμμα των αρμόδιων επιτροπών. Γι' αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε για τη δική μα γνωμοδότηση τον Οκτώβριο. Εξού και η πολύ σύντομη διορία για τι τροπολογίε. που λέγει όπως είπα στις 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι. Και λίγα λεπτά υπο, υπομονή, εν αναμονή του κυρίου Πιοτρόφσκη. We are waiting for the rapporteur. Actually for the rapporteurs. Περιμένουμε τον εισηγητή, μάλλον τους εισηγητές. Ούτε οι σκιώδεις εισηγητές. Ε, ή μάλλον ούτε οι εισηγητές στον επόμενο σημείο δεν είναι παρόντες για να περάσουμε σε άλλο θέμα. Okay, ladies and gentlemen, we can continue our... Μπορούμε να συνεχίσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή αυτή της συνεδρίασης. Περιμέναμε τον κύριο Πιοτρόφσκι, τον συντάκτη της γνωμοδότησής μας, που συμμετέχει, συμμετείχε σε συνεδρίαση σε άλλης επιτροπής, αλλά στο μεταξύ έχει έρθει και μπορούμε να συνεχίσουμε. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της της διάταξης, τη θέσπιση της διευκόλυνσης ή του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη. Εγώ σας παρουσίασα ήδη τη νέα πρόταση και σας ενημέρωσα για ποιες είναι οι καθα... κατ' ουσία αρμόδιες επιτροπές, οι επιτροπές βιομηχανίας, ήτρα και μεταφορών, τραν. Είναι συναρμόδιες δυνάμει του άρθρου 55 Σα είπα ότι αρμόδιος συντάκτης γνωμοδότης εκ μέρους της Επιτροπής είναι ο κ. και από το ECR και επίση υπενθύμησα ότι η διορία για τι τροπολογίε λήγει το μεσημέρι της Παρασκευής 7 ε, Σεπτεμβρίου. Και τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο και Σα ακούμε κύριε εισηγητά. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα την γραμματεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη συνεργασία που είχα εν ώψη της σύνταξης της έκθεσης, της γνωμοδότησης αυτής που αφορά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη που στα πλαίσια των διευρωπαϊκών προγραμμάτων, δικτύων μάλλον ε, μεταφορών, ε, θεωρεί ότι οδηγεί μια Ευρώπη προς με μηδέν νεκρούς, μηδέν εκπομπές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και επίσης με μια πρωτοπόρα ψηφιακή οικονομία. Επίσης θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τον άνθρακα, θέλουμε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και το συνδέοντα στην Ευρώπη θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε και αυτό το στόχο. Επίσης, ε, φυστώ την προσοχή σας στην ανάγκη χρηματοδότησης ε, των εσωτερικών πλωτών οδών, που είναι σημαντική οδή μεταφοράς. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα λοιπόν στις εσωτερικές πλωτές οδούς, αλλά και στα διασυνοριακά τμήματα των εσωτερικών πλωτών οδών, αλλά και ε, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και στις παραμεθόριες περιοχές. Ε, με βάση τις προ... πληροφορίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό. θα πρέπει να στηριχθεί σε ευιστάμενα κονδύλια και κυρίως σε ένα τμήμα των κονδύλιων της του Ταμείου Συνοχής. Πολλά όμως κράτη-μέλη ήδη έχουν δηλώσει την αντίθεση τους ε, απέναντι στην υπερβολική συρρήκνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής. Και συμφωνώ και εγώ με αυτή την ε, άποψη και την προσυπογράφω και την παρουσιάζω και στην γνωμοδότηση. Στην Επιτροπή Μεταφορών άκουσα ότι το θέμα της, ε, του Ταμείου Συνοχής δεν έχει οριστικοποιηθεί. Έγινε συζήτηση με τον επρόσωπο του ΕΛΚ και με τον κύριο Τελίσκα από το Σοσιαλιστή. Δεν έχει προεξοφληθεί λοιπόν το θέμα του Ταμείου Συνοχής. Μπορεί να αλλάξει. Είναι ακόμη ρευστό και ανοιχτό το θέμα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί και εγώ περιμένω τις δικές σας προτάσεις και τα σχόλιά σας που θα προσπαθήσω να τα λάβω υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε με τους σκιώδεις ηγετές. Κυρία Σμιτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είμαι μέλος της Επιτροπής Τραν ως ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για κάποια θέματα που αναφέρει ο εισηγητής θέλω να τα τονίσω και εγώ. Πρώτα, όπως είπε ήδη, την στόχευση στην υγροποίηση του άνθρακα, ως, δηλαδή του διοξιδίου του άνθρακος. Γνωρίζουμε ότι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως Audi και άλλες κάνουν ήδη σχετικά πειράματα. Η δε εταιρεία Shell άνοιξε ήδη το πρώτο μεγάλο διληστήριο για σχετικά καύσιμα, δυστυχώς όχι στην Ευρώπη, αλλά στο Κατάρ. Η τεχνολογία αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει τεράστιο δυναμικό ιδίω όταν πρόκειται για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακου στην ατμόσφαιρα. Σημαντικό επίσης το δυναμικό για την μείωση της γεωστρατηγικής μας εξάρτησης από χώρες που παράγουν ορυκτά καύσιμα. Και πρέπει να είναι στόχος του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ισχύει και ο δεύτερος χαρακτήρα τη τεχνολογία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να βασιστεί η Ευρώπη σε μια τεχνολογία, γιατί και σε κάθε χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορετικοί ε, πόροι ενέργειας. Άλλο στη Σουηδία, άλλο στην Πολωνία, άλλο σε χώρες του Νότου. Είναι σημαντικό, όπω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 30% των ε, κονδυλίων της ΕΦ να ανοίξουν στον ανταγωνισμό. Ω μέλος τη Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού θα παζητήσω 100% αλλά έχοντας υπόψη και τις μελέτες για την ανάπτυξη των ε, σχεδίων των σιδηροδρομικών δικτύων, έχω δηλαδή υπόψη μου και αυτό, εν ώψη τώρα της αναγκαία χρηματοδότησης και το πόσο περιορισμένα είναι τα κονδύλια της ΣΕΦ, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα κονδύλια αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της προβάλλει το θέμα της συνοχής και μέσα στα πλαίσια της ε, διευκόνησης συνδέοντας δηλαδή στην Ευρώπη. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις άλλες τροπολογίες που θα κατατεθούν έως τέλος της εβδομάδας. Το μήνυμα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ασφαλώς θα έχει σημασία πέραν των ορίων της γνωμοδότησης. Ένα τρίτο σχόλιο, όπως είδαμε στην προηγούμενη περίοδο, η Διευκόν συνδέοντα της Ευρώπης χρησιμοποιείται συχνά για άντληση κονδυλίων όταν τα έχει ανάγκη αλλού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν μπορεί να είναι σωστή βάση για την σωστή διαχείρισή της. Άλλωστε, ο τομέας των μεταφορών οφείλει να συμβάλλει σημαντικά για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακου, ταυτόχρονα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στη βάση ευθυνών, οικονομικών δηλαδή, μεταφορών. Θα κάνω σχετικές τροπολογίες που θα περιλαμβάνουν πιθανώς και αύξηση της χρηματοδότησης για την διευκόλυνση γενικά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Ροντρίγκε που εκπροσωπείται τον κύριο Μποστινάρου, ή μάλλον η κυρία Ροντρίγκε, με συγχωρείτε, εκπροσωπεί τον κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Δυστυχώ ο κύριο Μποστινάρου δεν μπόρεσε να προσέλθει. Έχω λίγα λόγια να πω λοιπόν στο όνομά του. Πρώτα ο κ. Μποστινάρου τονίζει τη σημασία της διευκόνησης συνδέοντα στην Ευρώπη και τη σχέση μεταξύ αυτής και του Ταμείου Συνοχής. Όταν άρχισε πριν ε, από μια εξαετία η συζήτηση για την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη, η συζήτηση να μεταφερθούν κάποια κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής στην ΣΕΦ είχε εμφανιστεί ως ένας τρόπος για να καλυφθούν κάποια κενά στο, δίκτυο των τεντή, Το γεγονός ότι παραμένει η πρόταση αυτή μεταφοράς και στη νέα πρόταση και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, αν δούμε δηλαδή τα νούμερα σχετικά, μειώνονται τα κοντήρια του Ταμείου Συνοχής στο μισό. Ενώ παραμένει αναλύωτη η συμβολή του στην ΣΕΦ. Αυτό πρέπει να συζητηθεί. Κάτι που πρέπει να συζητηθεί όμως το επίπεδο του CPR, όχι του κανονισμού για την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Θα κάνει σχετικέ προτάσει ο κ. Μποστινάρου, όπως είχε γίνει και προεξέτηες να μην αναφερθούν δηλαδή νούμερα συγκεκριμένα τώρα για την μετακίνηση κοντιλίων από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό θα πρέπει να μείνει κενό. Και οι διαπραγματεύσει CPR θα πρέπει να στραφούν γύρω από το αν θα διατηρηθεί η μεταφορά αυτή και τελικώ και το ποσό. Ο κύριος Μποστινάρου θα παρέμβει και στο άρθρο 4.8 για την χρήση που μπορεί να γίνει των κονδυλίων που θα μεταφερθούν από το Ταμείο Συνοχής. Προεξαετίας ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο το θέμα αυτό, διότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προσέφερε εγγύηση στις χώρες της συνοχής ότι τα χρήματα που μετέφερε κάθε μια από αυτές στο ΣΕΦ θα χρησιμοποιούνταν για ολοκλήρωση έργων στην ίδια τη χώρα μέλος. Το πρόβλημα προέρχεται από το ότι το Ταμείο Συνοχής έχει επιμερισμένη διαχείριση, ενώ η ΣΕΦ είναι σε, συγκε... σε κεντρική διαχείριση. Ο κ. Μποστινάρου ήταν επίση εισηγητή για τον κανονισμό του Ταμείου Συνοχή και τότε είχε επιτευχθεί μια σημαντική συμβαστική λύση. Για τα πρώτα τρία έτη δηλαδή τη εφαρμογή, η μεταφορά κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχή στην ΣΕΦ μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά μόνο στην ίδια αυτή τη συγκεκριμένη χώρα μέλο που έκανε τη μεταφορά. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή και δεν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση που γίνεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρηθούν μόνο 70% των πόρων η ρήτρα διαφύλαξη που είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη φορά πρέπει να παραμείνει και να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή των εθνικών αυτών συνεισφορών. Πρέπει να γίνει πρόοδος για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν Όλοι οι πόροι μεταφέρονται στην ΣΕΦ. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί τεχνική ενίσχυση, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, και να προσθεθούν όσο γίνεται περισσότερο οι διοικητικέ διαδικασίε. Σε ό,τι αφορά τι προτάσει του εισηγητού, ο κ. Ποστινάρου βρίσκει ότι υπάρχουν προβλήματα με την διαγραφή της λέξης decarbonization και ταυτόχρονα για τη σχετική τεχνολογία. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της ρήπανση. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια τελική καθαρή λύση. Τέλος, το μήνυμα του κ. Ποστινάρου είναι ότι θα καταθέσει κάποιες τροπολογίες στην κατεύθυνση αυτή με τα μηνύματα που μόλις σας ανέβηξα εκ μέρους του. Ευχαριστώ πολύ. να να παραστεί ως και ο Θέλω να πω ότι με χαροποιεί η τελευταία παρατήρηση με κλίση το γεγονός ότι ε, μιλάμε για decarbonization, σαν να μην υπήρχε η Συμφωνία των Παρισίων. Πραγματικά με πλήση το να βλέπω ότι μιλάμε για τεχνολογία καθαρού αρτρακά. Μιλάμε για επένδυση στις υποδομές και οι υποδομές θα πρέπει να μας παρέχουν την δυνατότητα βιώσιμης μετακίνησης. Ενδεχομένως υπάρχουν τα συμφέροντα της Πολωνίας. Κατά την άποψή μου όμως δεν είναι σωστό αυτό. Εδώ μιλάμε για ένα κεφάλαιο που είναι σημαντικό για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τις μεμονωμένες χώρες. Τροπολογία 8 η αγορά κονδυλίων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις ενισχύσεις. Όχι, πρόκειται για μια χρηματοδότηση της εθνικής πολιτικής ε, με ευρωπαϊκά κονδύλια. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να καθορίσουμε τις προστιθέμενες αξίες. Συχνά αυτό έχει σχέση με πολιτικές φίλων των κρατών. Εγώ δεν θα ακολουθούσα αυτόν τον δρόμο. Θα με φόβιζαν οι εκθέσεις της Όλαφ και του Ελεκτικού Συνεδρίου σε μερικά χρόνια. Με η αναφορά στις άκρος απομακρυσμένες περιοχές έχει ε, αφαιρεθεί. Εγώ είμαι πολιτικός που ενδιαφέρομαι και την Ευρώπη. Υπάρχουν τέτοιου είδους περιοχές που θα πρέπει να συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη και θα πρέπει να συνδέονται και με τις κοντινές περιοχές. Μου θυμίζει, ε, ε, είναι κάτι ε, πολωνέζικα αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Τελευταίο σημείο. Πολύ συχνά στην Επιτροπή Μεταφορών κάνουμε αναφορά για το πώς θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους μας δαπανώντας ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί και με την πραγματοποίηση διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενδεχομένως με το Connecting Europe Facility. Αυτό που κάνουμε τώρα στο αμείο συνοχή θα μπορούσε να γίνει και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό συνδέεται με σημαντικά θέματα που αφορούν περιοχές πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα δηλαδή του διευρωπαϊκού δικτύου. Τα χρήματα δεν θα πρέπει να δοθούν μόνο για το ε, δίκτυο πυρήνα, αλλά για ένα παγκόσμιο δίκτυο, που είναι σημαντικό σε επίπεδο περιφερειακό. Θα ήθελα να σας προτείνω σήμερα αυτή την ιδέα, θα υποβάλω και μία ε, ε, τροπολογία. Ήθελα όμως να ρίξω τώρα την ιδέα και να μιλήσω υπέρ αυτής γιατί το ίδιο ευρώ που δαπανάται στην Ευρώπη θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίτευξη περισσότερων στόχων. Δεν βλέπω τον κύριο Ράγκμουν. Άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Σόρμπιχτ. Ευχαριστώ. Ε, Σύντομε παρατηρήσει, αν μου επιτρέπετε. Η πρόταση του κυρίου Μποστινάρο να παραμείνει κενό ότι ε, όλες οι επιτροπές ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση. Και στην Επιτροπή Προπολογισμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα εθνικά κονδύλια στον πρώτο γύρο και τώρα προσπαθούμε να προετοιμαστούμε στην ενδιάμεση έκθεση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, θα θέλαμε οι επιμέρου επιτροπέ συμπεριλαμβανομένε και τη δική μα να εκπονήσουν τι προτάσει του για τα συγκεκριμένα κονδύλια και να προτείνουν συγκεκριμένα ποσά. Και αυτό θα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο ως πρώτη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα είναι κενό το σημείο αυτό. Θα είναι με συγκεκριμένα ποσά, με νούμερα. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούσαμε ότι το Ταμείο Συνοχής καλύπτει με διάφορους τρόπους. Αυτή είναι η, ε, επιμερισμένη διαχείριση. Από τη στιγμή όμως που έχουμε άλλου είδους ε, διαχείριση, δεν είναι μόνο η μέθοδος που αλλάζει, είναι το είδος της διαχείρισης αλλάζει. Και από τη στιγμή που θα αναλάβουν τα κράτη-μέλη, ε, από τα εθνικά τους κονδύλια, αυτά λειτουργήσαν καλά αλλά δεν ήταν αυτό που είχε είχαν υποσχεθεί για την συνοχή. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε περικοπή του Ταμείου Συνοχής κατά 40%. Είπε να επιστρέψουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα φυσικά επίπεδα. Όμως μειώνεται το Ταμείο Συνοχής, ο προϋπολογισμός του. Και το συνδυάζουμε με, το με τη διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι ότι έχουν παραμείνει άθικτα τα κονδύλια. Είναι και έχουμε λιγότερα κονδύλια στη συνοχή και μερικά μεταφέρονται στη, στο συνδέοντα στην Ευρώπη. Επίση ό,τι αφορά τον καθαρό άνθρακα. Αντιλαμβάνομαι ότι ιδεολογικά η ιδέα του καθαρού άνθρακα αντιβαίνει στην ε, Συμφωνία των Παρισίων, αλλά θα σα δώσω το παράδειγμα του Ελσίνκη, ε, που χρησιμοποιεί άνθρακα για τη θέρμασή του. Οπότε α είμαστε λίγο πιο σοβαροί και θα πρέπει να σκεφτόμαστε που και που και νέε τεχνολογίε, ιδιαίτερα σε χώρε που έχουν μια οικονομία που στηρίζεται στον άνθρακα. Α μην το απορρίψουμε λοιπόν αμέσω με μια μονοκονδυλιά το θέμα του άνθρακα με πρόσχημα την Συμφωνία των Παρισίων. Υπάρχουν δυνατότητε και όντω καθαρών τεχνολογιών άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, ο κύριο Βανίστερο. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντα τον ηρμό του προηγούμενου ομιλητή. Το έχουμε ξανασυζητήσει και το είχαμε πει και πέρυσι. Θα έχουμε ένα, ποσοστό, ένα ποσό για τις μεταφορές ή ένα δίκαιο μερίδιο. Γιατί όταν ε, ε, έχουμε, έχει περιοριστεί η, η τούρτα, δεν μπορούμε να κρατήσουμε ε, τα μεγάλα κομμάτια της προηγούμενης τούρτας. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες διαστάσεις. Και αυτό το δεχτήκαμε και στην Επιτροπή και στην ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά μερικές φορές τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν πώς να εναρχίζουν τις προτεραιότητες τους. Και καμιά φορά θα πρέπει να ρίχνουν μια ματιά και στις γειτονικέ τους χώρες. Και ξέρουμε ότι στη δεύτερη περίοδο προγραμματισμού θα γίνει κεντρική διαχείριση, οπότε μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Γίνεται ένα συνδυασμό των δύο συστημάτων δηλαδή. Και Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον παράγοντα χρόνο. Αλλά ίσως δεν γίνει καν συζήτηση για το άδικο μερίδιο. Οπότε τότε είναι που θα εξεγερθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση μου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όντως. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή και τους ε, σκιώδη ηγητές και τους υπόλοιπους ομιλητές. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το θέμα του κλίματος. Ξέρετε ότι προτείνουμε 25% του μακροπρόθεσμου συνολικού προϋπολογισμού να αφορά το κλίμα και το συνδέοντα στην Ευρώπη έχει ένα σημαντικό μερίδιο αυτού. Προτείνουμε στόχο 60% για το ε, ΣΕΦ γενικά για τους τρεις τομείς. Οπότε συμφωνώ με τα σχόλια ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τη μνήα της απαλλαγής από τις εκπομπές άθρακα και δεν μπορούμε να δεχτούμε τον καθαρό άθρακα γιατί το συνδέοντας στην Ευρώπη δεν χρηματοδοτεί παραγωγή ενέργειας, αλλά επικεντρώνεται στην μεταφορά ενέργειας. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το κονδύλιο της συνοχής. Το τρέχον κονδύλιο της συνοχής έχει λειτουργήσει θαυμάσια και μάλιστα έχει απορροφηθεί πλήρως, έχει εκταμιευθεί πλήρως τη στιγμή που μιλάμε. Όλα τα κρατημέλη ε, χρησιμοποίησαν σχεδόν στο έπακρο με μία μικρή διαφορά. Μόνο δύο χώρες ε, και με λίγα εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να εκμεταμιεύσουν πλήρως τον εθνικό του κονδύλιο και τώρα βλέπουμε την πρόοδο στις διάφορες δράσεις. Και εφαρμόζουμε την αρχή use it or lose it ή το χρησιμοποιείς το χάνεις και για μερικά προγράμματα που δεν λειτουργούσαν θα ξαναμπούν στον κορβανά και θα αναδιανεμηθούν. Φυσικά μόνο μεταξύ των χωρών της συνοχής. Και θέλουμε να διαφυλάξουμε αυτή την αρχή και τον κανόνα των τριών ετών και την αρχή του use it or lose it. Το θέμα είναι ότι ένα μικρό κλάσμα αυτού του κονδυλίου θα υπόκειται στον ανταγωνισμό από την αρχή. Και γιατί το προτείνουμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα του κονδυλίου που καθορίζουμε, αλλά θέλουμε αυτό το κονδύλιο να χρηματοδοτεί διασυνοριακά προγράμματα και η ιδέα των εθνικών κονδυλίων συνδέεται κυρίως με εθνικά προγράμματα. Αν όμω ένα μικρό τμήμα το εντάξουμε στον ανταγωνισμό και αφήσουμε να παίξει ο ανταγωνισμό, θα προσανατολίσουμε καλύτερα ένα τμήμα του κονδυλίου στα διασυνοριακά σχέδια. Επίση, ο γενικό ε, προπολογισμό, το γενικό κονδύλιο του Συνδέοντα στην Ευρώπη, ε, τα κυρώνεται με βάση την ανταγωνιστική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ξέρετε ότι θέλαμε η ρητή μνήα στον κανονισμό του ιδιαίτερα στην Ευρώπη για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές προκειμένου να συμμετέχουν στα προγράμματα, γιατί μέχρι στιγμής δεν συμμετείχαν ε, σε επαρκές επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν ρητή μνήα των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να τους επιτρέψουμε να λάβουν μέρος και μα προβληματίζει ιδιαίτερα η πρόταση να αφαιρεθεί η ρηφή αυτή η μνήμα των εξόχων απόκεντρων περιοχών. Διαφωνούμε. Θέλουμε να παραμείνει αυτή η μνήμα για να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικέ ανάγκε των εξόχων απόκεντρων περιοχών σε ε, υποδομέ μεταφορών. Σα ευχαριστώ κύριε Πιοτρόφσκι. Θέλετε να δευτερολογήσετε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα, σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα του συναδέλφου ε, που ε, έλαβαν το λόγο, σημείωσα διεξοδικά τα σχόλιά τους και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη στη συνέχεια ε, τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές ε, προτάσεις. Και μάλιστα το τελευταίο σχόλιο τη Επιτροπή για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ ε, το λαμβάνω υπόψη και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβασμό και για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ, αλλά και τις παραμεθόριες περιοχές Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωσης. Ε, και ευελπιστώ ότι και για άλλα σημεία θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στη συζήτηση και για τα σχόλιά σα. Μάλιστα, να σα υπενθυμίσω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 12. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης που είναι η ενδιάμεση έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την περίοδο 2021-2027. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη συμφωνίας. Η συγητής μας για την γνωμοδότηση είναι ο κύριος Ντέρεκ Βόν, Αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έχουμε τέσσερις εισηγητές ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, συνεισηγητές για το θέμα αυτό και ο κύριος Όλμπριχτ είναι ένας από αυτούς τους τέσσερις και ελπίζουμε ότι θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση 8 ή 9 Οκτωβρίου γι' αυτό και ορίσαμε την ε, διορία και τις τροπολογίες μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βόν για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ξέρετε ότι προβλέπεται η υπηρεσία συνένεσης και αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προπολογισμού να συντάξει μία προσωρινή έκθεση έτσι ώστε θα μπορεί να μπορέσουν να προβληθούν όλα τα επιχειρήματα και αυτό κάνει τη ζωή ευκολότερη για το Γιάννη. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της γνωμοδότησής μου, αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να κάνω μια αναφορά στη θέση του Κοινοβουλίου που θα υιοθετηθεί το Μάρτιο. Δηλαδή, ε, είπα ότι θα πρέπει να διατηρηθούμε στο πλαίσιο του 3,5 σε ό,τι αφορά τις διαδροτικές πολιτικές και την παρούσα περίοδο του ε, προϋπολογισμού. Και να έχουμε την βεβαιότητα ότι γίνονται σεβαστές οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Συνοχής, σύμφωνα με την πρόταση του Κοινοβουλίου, θα είναι 272 δισεκατομμύρια ευρώ που θα ε, μοιραστούν μεταξύ του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Η Επιτροπή έκανε αυτό τον διαχωρισμό και γι' αυτό το λόγο αναφερόμαστε και εμείς αυτό. Επιβεβαιώνω ότι η Επιτροπή Προεπροϊσμού πιστεύει ότι θα πρέπει ε, να συζητηθεί περαιτέρω αυτό το θέμα. Οι συνάδελφοι βεβαίως μπορούν να υποβάλουν πρωτοβουλίες, ε, ε τροπολογίες, αποφασίσουν πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Εξετάσαμε επίσης το χαρτοφυλάκιο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κρατήσαμε τις ε, πιστώσεις οι περισσότεροι συνάδελφοι θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερθήκαμε και στο θέμα του Ίντερεγκ. Η Επιτροπή αναφέρεται στο 2,7%. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ένα νέο πρόγραμμα το οποίο προκάλεσε πάρα πολλές ε, συζητήσεις και σε αυτήν την Επιτροπή και σε άλλες Επιτροπές. Οι συνάδελφοι σας γνωρίζουν την πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα καινούριο ε, εργαλείο. Κατά την άποψή μου, τα περισσότερα κονδύλια θα μπορούσαν να να δαπανηθούν καλύτερα κάπου αλλού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ιντερεκ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό είναι το ερώτημα για τους ε, συναδέλφους. Είπαμε ότι πραγματικά αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα προς ε, συζήτηση. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψη των συναδέλφων για αυτό το θέμα. Τέλος, ε, κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την άποψη που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο, προτείνω να περάσουμε από τα 600 εκατομμύρια στο 1 δίσα. Αυτή ήταν η θέση του Κοινοβουλίου φέτος ε, το Μάρτιο. Όπως ε, ε, είπατε, το, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι ειδικά τη Σεπτεμβρίου. Thank you, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βόν. Τώρα, σκιώδεις συγητές. Ε, είναι περιορισμένε κάπως οι πληροφορίε μου, γι' αυτό για παρακαλώ να με διαφωτίσετε. Ποιος θα λάβει το λόγο εκ μέρου του Λαϊκού κόμματο. <laughs> για να σα βοηθήσω κυρία Πρόεδρε να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Ο μεγάλο συνάδελφό μου, ο κύριος Σιλό είναι... Ζουλό. Ζουλό. Αλλά ε, δεν ε, έχω το κείμενό του, παρά μόνο στα γαλλικά. Τώρα, να μιλήσω, να πω στον εισηγητή, διότι κάποιος ο οποίος είναι πλησίον της πραγματικότητας και γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, αυτός είναι ο κύριος Βόν. Διότι επί χρόνια είναι μέλος της Επιτροπής Προπολογισμών και βεβαίως και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και αυτή είναι, αυτός είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Αν δείτε καλά τη γνωμοδότησή του, θα δείτε ότι έχει περιλάβει τα πάντα και τι έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο ως δικές του επιθυμίες. Και τα πραγματικά νούμερα. Εκεί έχουμε την ίδια προσέγγιση. Και προωθεί επίσης και την αναγκαιότητα να μην γίνεται διάκριση ανάμεσα στην απόδοση κάποιων παραδοσιακών πολιτικών και στι αλλαγέ που γίνονται. Δεν υπάρχουν απειχιωμένε παραδοσιακέ πολιτικέ Πρόκειται για πολιτική συνοχή η οποία πράγματι ακόμη αποδίδει. Αλλά χρειάζεται κάποιε αλλαγέ. Αυτό είναι το σωστό. Και εδώ το λέει αυτό και ο κύριο Ζουλό. Επίση το γεγονό ότι έγινε μια συζήτηση και ο κύριο Ζουλό έχει συντάξει την έκθεσή του για την 7η έκθεση συνοχή την οποία στην οποία δείξαμε με νούμερα ποια ήταν η συμβολή στην προστιθέμενη αξία και στο πρασίνισμα της Ευρώπης και στην ευφιέστερη Ευρώπη και σε μια Ευρώπη ανάπτυξης και απασχόλησης. Υποστηρίζει ο κ. Ζουλό λοιπόν το βασικό μήνυμα στην έκθεση του κ. Βον, στην γνωμοδότηση του κ. Βον, επικρίνει τις ε, βαριές περικοπές στο Ταμείο Συνοχής Ιδίω. Αυτή είναι η γενική γραμμή του κ. Ζουλό. Σήμερα συζητήσαμε το πρώτο σχέδιο της έκθεσης Interreg επίσης και είδαμε ότι είναι και αναγκαίο να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για το Interreg και εκεί συμφωνήσαμε όλοι. Υπάρχει λοιπόν μια καλή βάση. Ο κ. Ζουλό θα πράξει πάντο δυνατό για να καταθέσει και σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ, λέει ο κ. Βανίστερο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από ECR δεν έχουμε. Άλντε η κυρία Κατάινεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον εισηγητή, κύριο Βόν. Πράγματι η δουλειά που έχει κάνει είναι εξαιρετική. Έχω συνεργαστεί και στην Επιτροπή Προεπολισμών με τον κύριο Βόν και βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Και συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπέ στο πρόγραμμα Interreg. Και συμφωνώ επίση ότι πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της ανακαίνησης κτηρίων και να δοθούν χρήματα σχετικά. Αυτά και στα πλαίσια της προώθησης μιας βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα και με τους στόχους της χιλιετίας των ΗΕ. Και εκεί είναι πολύ σημαντική και η διάσταση του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ με τη σειρά μου τον κύριο Βόν που έχει περιλάβει στη γνωμοδότησή του πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία ε, στηρίζονται και θεμελιώνονται και σε στατιστικές και βεβαίως και με ποσοστίες αναλογίες κλπ. Εάν μπορέσουμε να επιβάλλουμε τις προτάσεις αυτές, το κείμενο τελικό θα είναι πάρα πολύ θετικό. Και ελπίζω να αποτελέσει ένα σημαντικό άλμα στην πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, πάντως, να Υποβάλλω και κάποιες άλλες ιδέες. Γνωρίζω ότι είναι παρόν η παρούσα η εκπρόσωπος της Κομισιόν και θα μπορέσει να τα σημειώσει. Πρόκειται για τις πολιτικές προς όλες τις ε, περιφέρειες. Η Λιθουανία, νομίζω και άλλες χώρες, το 2016 είχε λάβει απόφαση να τροποποιήσει την πολιτική της, να μην είναι δηλαδή πλέον ενιαία περιφέρεια και να ασκήσει πολιτικές κομμένες και ραμμένες για διαφορετικές περιφέρειες μέσα στην ίδια την χώρα. Το 2017 την απόφαση αυτή τη στήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2018 προέκυψε νέα κατανομή περιφερειών, ωστόσο οι προτάσεις που κατατέθηκαν έγιναν πάλι στην βάση της παλαιάς περιφερειακής η οποία δεν ισχύει πλέον σήμερα. Γι' αυτό θα καταθέσω μια σχετική τροπολογία σχετικά με τη νέα περιφερειακή κατανομή. Υπάρχουν ε, δύο περιφέρειες που προέκυψαν το 2017. Δεν υπήρχαν το 2016. Πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές, διότι αν ληφθούν όλα τα μέτρα στην βάση μια ενιαία περιφέρεια που συμπίπτει με την επικράτεια δηλαδή, δεν θα προκύψει το υποθεμένο αποτέλεσμα. Ελπίζω να μπορέσει ε, να δείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναγκαία ευελιξία και να λάβει υπόψη τις περιφέρειες αυτές, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι αποφάσεις που έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ε, δύο νέων περιφερειών στηρίζω τις προτάσεις του Γρυβών σε ό,τι αφορά τη συνοχή. καθώς και την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, ο κύριος Βαν Μίλτενμπεργκ. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Πολύ σύντομα ομιλώ εξ ονόματος μέρους των φιλελευθέρων, μιλώντας για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ρεαλισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην εμείνει σε μια πολιτική να αντιληφθεί ότι το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο οφείλει να αρθεί στο ύψο των σημερινών προκλήσεων που είναι πολύ διαφορετικέ από αυτέ που ήταν πριν από 7 ή 10 χρόνια. Πρέπει να δεχθούμε ότι θα ε, είναι αναγκαίο να γίνουν προσαρμογέ. και ίσω, να μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για το γεγονό ότι παρέμειναν οι περικοπέ κάπω περιορισμένε, χώρε όπως Πολωνία και Ουγγαρία έχουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι λογικό λοιπόν να λάβουν λιγότερα κονδύλια από τα Ταμείο Συνοχής. Μιλήσαμε πριν για τη συμβολή του Ταμείου Συνοχής στην διευκόλυνση της Ευρώπη. Αυτά πρέπει να περιεχθούν στη γνωμοδότηση. Βλέπω όμως ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες δεν θέλουν να στηρίξουν καμία μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Μιλούμε όμως για τα χρήματα των φορολογουμένων και οφείλουμε να κάνουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις ώστε οι επενδύσει όταν γίνονται να οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα. Θα είναι μια χαμένη ευκαιρία εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεχθεί την άποψη του εισηγητού. Εγώ τάσομαι υπέρ μιας ισχυρότερης στόχευσης σε κάποια σημαντικά θέματα στο μέλλον δηλαδή, για το μέλλον δηλαδή του Ταμείου Συνοχής. Σας ευχαριστώ κύριε Σόλμπριχτ. Ευχαριστώ. Να προσθέσω κάτι συμπληρώνοντα τον κύριο Βόν, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Να σε εξηγήσω την διαδικασία που πρότεινε η Επιτροπή Προπολογισμών σε σχέση με τη δική, σας επιτροπή, με τη δική μας επιτροπή, την Επιτροπή Ρέγγι και τις υπόλοιπες επιτροπές. Όπως είπε ο Τέρεκ Βον, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου ήταν 1,3 του ακαθάριστο χώριου εισοδήματο και αυτό θα, παρα... θα το κρατήσουμε. Σε αυτό θα εμείνουμε, στο ποσοστό 1,3 του GNI. Δεν θα είναι εύκολο γιατί μερικές επιτροπές θα ήθελαν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δίνεται να είναι πιο απαιτητικό, γιατί τα κράτη-μέλη ουδέποτε δεν θα συμφωνήσουν σε ένα υψηλότερο ποσοστό από το 1,3. Ακόμη και το 1,3 για πολλά κράτη-μέλη είναι υπερβολικό και αδύνατο. Θα πρέπει όμως να είμαστε συνεπείς και να εμείνουμε στο 1,3 ως ανώτατο όριο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που προτείναμε και το ψηφίσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την πολιτική συνοχής στο ονομαστικό επίπεδο του 2018. Το σημερινό δηλαδή επίπεδο τη ονομαστική αξία. Αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή είναι η λιμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε το θέμα είναι πώς θα μεταφέρουμε ε, αυτή την απόφαση και στο αριθμητικό επίπεδο. Ο προκαταρκτικός ε, πίνακας με τα ποσά, με, τους, ε, τα νούμερα, είναι, θα πρέπει να απόρρια αυτή τη απόφαση. Οπότε θα πρέπει να δούμε σε Επιτροπή Προπολογισμού τι θα σημαίνει να το κρατήσουμε στα επίπεδα τα σημερινά τα ονομαστικά. Δεν μπορούμε όμω, η Επιτροπή Προπολογισμού δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Επιτροπή Ρέγγι στι συζητήσει για τα ταμεία. Δεν μπορεί η Επιτροπή Προπολογισμού να συζητήσει ποιο ταμείο θα έχει περισσότερα κονδύλια και πιο λιγότερα. Εμεί κρατάμε το γενικό κονδύλιο τη συνοχή και περιμένουμε ε, από τον συντάκτη της γνωμοδότησης Επιτροπής Ρέγγι να πει ότι η Ρέγγι θεωρεί ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος ε, για να σεβαστούμε το γενικό κονδύλιο που είναι το όριο που έχει ήδη αποφασιστεί. Οπότε αυτή είναι η πολιτική ε, διάσταση μεταξύ των τριών ταμείων του Περιφερειακής Ανάπτυξης, ε, του Ταμείου Συνοχής και του ενισχυμένου ΕΚΤ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό όμω δεν θα το κάνει η Επιτροπή Προπολογισμών, γιατί αν μπούμε σε λεπτομέρειε, θα πρέπει η Επιτροπή Προπολογισμών να αποφασίσει για τη Γεωργία για τον ορίζοντα 2020. Όχι, εμεί είπαμε να κρατήσουμε το 1,3, να εμείνουμε στην απόφαση για το 1,3 και το Γενικό Κονδύλιο γιατί τα επιμέρους σημεία και την ανακατάταξη θα τα βρουν οι επιτροπέ. Αυτό αποφασίσαμε και με τον Ντέρεκ και θα θέλαμε εμείς στην Επιτροπή ε, προϋπολογισμών να ψηφίσουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στην Ολομέλεια. Και αυτή θα είναι η πολιτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν συνεχεία θα περιμένουμε τη θέση του Συμβουλίου. Και αυτό είναι πολύ ε, αβέβαιο, αν θα καταλήξει κοινή θέση το Συμβούλιο. Το θέμα είναι, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε αποκρισταλώσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο. Οπότε, η θέση του κυρίου Βον δεν είναι γενική, να είμαστε όλοι υγιείς και πλούσιοι, αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα επιμέρους σημεία. Ευχαριστώ κύριε Όλμπριχτ και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βον και συμφωνώ με τα σχόλιά του ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και δικό μας ε, συντάκτη γνωμοδότηση και δική μας γνωμοδότηση όπως έχουμε ε, ως, ξεχωριστή γνωμοδότηση του, της Ρέγγι. Ε, για ποια ολομέλεια του Νοεμβρίου ε, στην αρχή την πρώτη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τον Οκτώβριο θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει για το Brexit. Οπότε είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Πάντως μέχρι στιγμής το Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποβάλει την πρότασή του για το 1,3 το Νοέμβριο. Αυτή είναι η πολιτική απόφαση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο τι θέλει το Συμβούλιο και ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου ενδεχομένω. Μάλιστα, καλώ. Τώρα περνάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γέλα, να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω και κυρίω το συντάκτη τη γνωμοδότηση αλλά και την Επιτροπή γενικώ για του ταχύ ρυθμού με του οποίου κηρυθήκατε. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε στη συμφωνία για τα βασικά στοιχεία του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι την άνοιξη του χρόνου. Κατέγραψα τη θέση που προτείνεται για την πολιτική συνοχή γενικώ. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν διαφορετικά βασικά σενάρια και ξεκινούν από διαφορετικά σημεία. Και μάλιστα οι συζητήσει για αυτά τα σενάρια τα βασικά έγιναν αλλού Πάντως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Γενική Πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι πολύ ισορροπημένη για το συνολικό προπολογισμό και λαμβάνει υπόψη όλες τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριο Ροπέ έθεσε μια συγκεκριμένη ερώτηση για την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχουμε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο διαφορετικά στοιχεία. Έχουμε την περιφερειακή διάσταση σε σχέση με τη βάση υπολογισμού για την κατανομή των κονδυλίων και έχουμε την περιφερειακή διάσταση σε σχέση με τον προγραμματισμό και την οργάνωση των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση των προγραμμάτων, εκεί υπάρχει αρκετή ευελιξία, ελαστικότητα για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες που μπορούν να, οργανώσουν τη δομή των προγραμμάτων τους όπως θέλουν. Στο παρελθόν είχαμε μια γενική προσέγγιση ότι ο προγραμματισμός γίνεται σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Αλλά αυτό δεν ήταν απόλυτο κριτήριο. Και στα πλαίσια της διαδικασίας απλούστευσης για την επόμενη περίοδο έχουμε αφαιρέσει ακόμη και αυτό το σημείο αφετηρίας. Οπότε ε, ενισχύθηκε η ευελιξία για το πώς τα προγράμματα μπορούν και θα έπρεπε να οργανωθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βάση υπολογισμού για την κατανομή των κονδύλιων, εδώ έχουμε ένα απλούστατο στοιχείο. Για να έχουμε βάσει υπολογισμού για την κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ε, υπάρχουν εφόσον ε, οι περιφέρειες ε, έχουν θεσπιστεί για αρκετό καιρό ώστε να έχουν προλάβει να συγκεντρώσουν τα νέα στοιχεία. Οπότε, αν δεν έχουμε αυτή την προϋπόθεση, δεν θα έχουμε για πολλές ε, περιφέρειες ιστορικά στοιχεία για κατά τη στιγμή της ε, εφαρμογής της πρότασης. Τώρα, αυτό εξαρτάται από το πώς τα κράτη-μέλη δίνουν ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τις νέες κατηγορίες περιφερειών. Επίσης, η βάση για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπευλήθη το Μάιο ήταν τα τότε διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία την ημέρα τη υποβολή της πρότασης. Όταν έχουμε στατιστικά στοιχεία τα χρησιμοποιούμε, αλλά εδώ δεν είχαμε. Εξού λοιπόν η διαφορά μεταξύ των, της κατανομής των κονδύλων και του προγραμματισμού. Δύο επιπλέον τώρα σημεία που θα ήθελα να τονίσω από το σχέδιο γνωμοδότησης. Αναφέρθηκε επανειλημμένως η μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής. Και μάλιστα κάποιος ε, είπε ότι αφορά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μην έχουμε αυτή την ε, τεχνητή, αυτή διόγκωση του Ταμείου Συνοχής για τα νέα κράτη-μέλη που είχαμε στις δύο προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού. Και ε, ήταν τουλάχιστον ένα τρίτο του μεριδίου των χωρών για αυτές που μπήκαν μετά το 2004 και αυτό ήταν για να εξασφαλιστεί ένα, μια ελάχιστη κατανομή κονδυλίων για τις επενδύσεις ε, σε υποδομές μεταφορών και περιβάλλοντος. Τώρα, η προσέγγιση που υθετήσαμε μετά ε, για τις χώρες που έχουν πια πολιετή παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι αυτή η προσέγγιση δεν χρειάζεται πια ω θέμα τη μεθόδου κατανομή. Οπότε εφαρμόζουμε τη μέθοδο κατανομή πια άμεσα. Και το ποσό για το Ταμείο Συνοχή αφαιρείται από τη μέθοδο κατανομή και στη συνέχεια τα κράτη-μέλη κατανέμουν τα κονδύλια α, ανάλογα με τα ποσά. Δεν είναι ότι έχουμε, έχουμε περικόψει το Ταμείο Συνοχή, τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχή. Είναι απόρρια του υφιστάμενο τρόπου υπολογισμού που έχει πια, από, το οποίο, από τον οποίο έχει πια εκλείψει το ελάχιστο ποσοστό της κατανομής, το 1 τρίτο που υπήρχε πριν. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια για, τα, για τους συντελεστές συγχρηματοδότησης. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα και προηγουμένως στη συζήτηση για το Interreg. Όσο πιο ψηλό είναι το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο πιο χαμηλό είναι το συνολικό επενδυτικό πακέτο απλά και εξάστερα. Όσο περισσότερα απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερα από τα κράτη-μέλη, τόσο μικρότερος θα είναι ο γενικότερος προϋπολογισμός. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν θέτουμε ένα χαμηλότερο ποσοστό ε, συγχρηματοδότηση από αυτό που είχαμε στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Κύριε Βόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ φίλε και φίλοι για τις παρεμβάσεις σα. Νομίζω ότι γενικά είστε υπέρ τη ε, της γνωμοδότησης και ευχαριστώ ιδίω Βανίστερο και Κατάινεν. Έγιναν και προτάσει βεβαίω και σίγουρα θα κατεθούν και τροπολογίες στη γνωμοδότηση. Ίσως για τον προϋπολογισμό, ίσως για το CPR. Θα δούμε όταν θα έρθουν οι τροπολογίες. Για τον κύριο Βαν Μίλτενμπεργκ. Μιλεί για ορισμένα κονδύλια χωρών μελών. Δεν είμαι βέβαιος εάν εμείς ως Επιτροπή, ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή, μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για το εάν οι χώρες θα πρέπει να δεχθούν 10-15% περικοπές. Δεν νομίζω ότι αυτό εντάσσεται στην παρούσα γνωμοδότηση. Θα γίνει κάποια συζήτηση για το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γνωρίζω ότι τα υποστηρίζουν αυτά οι συναδελφοί μου. Και σίγουρα θα υποβληθούν τροπολογίες. Αυτό γνωρίζαμε από την αρχή. Είναι και από τα πιο δύσκολα ζητήματα που αντιμετωπίζαμε όταν συντάξαμε την γνωμοδότηση. Συμφωνώ με τον Γιάννη ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες, να λάβουμε κάποιες προτάσεις, κάποιες αποφάσεις, κάποιες ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα, κάποιες πολιτικές και ανάμεσα στο Ταμείο ERDF και στο Ταμείο Συνοχής για να δώσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μια γνωμοδότηση που να λέει τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει στη μεταρρύθμιση του Ταμείου. Είτε θα συμφωνήσουν οι συναδελφοί μου, είτε θα υποβάλουν τροπολογίες. Είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως για να συζητήσουμε και πριν από την εκπνοή της, της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών. Η πρόεδρος η οποία κατάθεση τροπολογιών είναι μέχρι στις 12 το μεσημέρι 10 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε το επόμενο θέμα πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεσή μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής με εισηγητή τον κύριο Κοζολίνο. Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής ε, πρόταση της 29ης Μαΐου και παρουσιάστηκε στις 20 Ιουνίου στην, ε, στην Επιτροπή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Κοζολίνο ορίστηκε εισηγητής. Την αρμοδιότητα επί της ουσίας έχει σε αυτό το θέμα η Επιτροπή Περιφερειακής Αναπτύξεως. Ο εισηγητής έχει συμμετάσχει ήδη, έχει οργανώσει ήδη κάποιες προπαρασκευαστικές συναντήσεις και τον ευχαριστώ. Σήμερα θα αναπτύξει τις πρώτες του σκέψεις για τον φάκελο και θα υποβάλει το σχέδιο της έκθεσής του 8 με 9 δεκάτου. Έχετε το λόγο κύριε Κοζολίνο για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως ε, η συζήτηση αυτή έχει σχέση με την ε, συζήτηση που κάνουμε. Η τελευταία συζήτηση είχε σχέση με τον ε, προϋπολογισμό. Το χρονοδιάγραμμά μας είναι αρκετά φιλόδοξο. Δηλαδή το να θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας μέχρι τον Νοέμβριο είναι πραγματικά ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Χρειάζεται βεβαίως και κάποια ταχύτητα που είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο το την επόμενη θητεία τους κανονισμούς και δεν τίθεται υπό συζήτηση η ποιότητα της εργασίας που θα πρέπει να επιτύχουμε και τα πολιτικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το πλαίσιο είναι γνωστό. Ο, παρα... ο κανονισμός για πρώτη φορά έχει λίγα άρθρα, αποτελεί μέρος μιας γενικότερης συζήτησης, στοχεύει ε, στο να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα κράτη-μέλη, υπάρχει μία ε, επικέντρωση στην ε, θεματολογία προκειμένου κατά κάποιον τρόπο να βοηθηθεί ένα ενιαίος προγραμματισμός των περιφερειακών ταμείων και πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό δεδομένο που προκύπτει από την ανάγνωση των διαφορών άρθρων. Μία εργασία ιδιαίτερα απλοποιημένη, λίγα άρθρα, αλλά ε, επικέντρωση σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτό μου φαίνεται κάτι θετικό, αλλά μας οθεί ε, να εργαστούμε επί το μεμονωμένο άρθρο. Τώρα, δεν θέλετε να επισέλθω θέματα ουσίας έγιναν ήδη συναντήσεις με την Επιτροπή, με τους συναδέλφους, με το σκιώδη συγητή, με τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να κάνω μια ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων. Καταρχάς, την πρόταση. Ξεκινάμε από το άρθρο 2. Εκεί που μας αναφέρει πέντε μικροπεριοχές, 21 τομείς ε, παρέμβασης. Ε, αυτό στο παρελθόν οι μακροπεριοχές ήταν 11. Εδώ ε, η προσοχή επικεντρώνεται σε 5 μικροπεριοχές και σε 21 τομείς παρέμβασης. Εδώ προστίθεται το άρθρο 3, όπου η, το θέμα της ευελιξίας των μεμονωμένων χωρών που έθιξα είναι ακόμα πιο σαφές. Εδώ υπάρχει μία συγκέντρωση θεμάτων σε εθνικό επίπεδο και μία ταξινόμηση η οποία γίνεται όχι χρησιμοποιώντας το ΕΠ σε περιφερειακό επίπεδο που συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά χρησιμοποιώντας προκειμένου να προωθηθεί αυτή η συγκέντρωση το ε, ε, το, το εισόδημα, το ακαθάριστο εισόδημα, γιατί και αυτό θέτει ορισμένα θέματα προς συζήτηση, όπως θα σας πω και αργότερα. Όχι μόνο δεν μας βοηθάει να δούμε τις διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων χωρών, αλλά δεν μας βοηθάει να δούμε τις διαφορές στις μεμονωμένες χώρες. Αυτό αφορά το άρθρο 3 σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, υπάρχει το θέμα της τεχνικής βοήθειας. Όπως ορίζεται. Θα ήθελα να ξεκινήσει εδώ μια συζήτηση. Είναι ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει με βάση την εμπειρία ε, που καταγράψαμε ενισχύοντας ιδιαίτερα τη δημόσια διοίκηση τα εργαλεία μέσω των οποίων προωθούμε την πολιτική συνοχή. Πώ δηλαδή η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε περαιτέρω να διευκολύνει αυτή την εμπειρία. Για παράδειγμα, στην Ιταλία υπάρχουν προγράμματα, ε, πολύ σημαντικά προγράμματα διοικητική ενίσχυση και για την Επιτροπή ήταν ένα σημείο καμπής. Συνεπώς θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή της τεχνικής βοήθειας ενισχύοντας τη διοικητική μηχανή. Το άρθρο 6 αφορά όλους τους τομείς που αποκλείονται από την ε, παρέμβαση του Ταμείου. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα επί των οποίων διεξάγεται μία συζήτηση. Μπορούμε, για παράδειγμα, να αποκλείσουμε ε, από τους κοινοτικούς, ε, την κοινωτική χρηματοδότηση, την πολιτική ε, συνοχή σε ό,τι αφορά τον κύκλο των ε, απορριμμάτων. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που θα πρέπει να διευκρινίσουμε, θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Τώρα, το άρθρο 7 με την ίδια την Επιτροπή αποφασίσαμε σε ό,τι αφορά τους δείκτες να σκεφτούμε περαιτέρω το θέμα και να ανταλλάξουμε απόψεις για να μπορέσουμε να δούμε διεξοδικότερα αυτά τα θέματα που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την επίπτωση που έχει η πολιτική συνοχής. Εγώ προσπάθησα να κάνω μία σύνθεση για να μην μακρηγορήσουμε ιδιαίτερα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία ενός κανονισμού που αποτελείται, είναι ευέλικτος, αποτελείται από λίγα άθρα, αλλά μας ε, επιβάλλει να εργαστούμε προσεκτικά. Το θέμα του Ταμείου Συνοχής που αφορά τις περιφέρειες και το θέμα των πόρων, όπως είπαμε και προηγουμένως, παραμένει ένα θέμα εκρεμέσα. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα περαιτέρω. Δύο παρατηρήσεις ο γενικού χαρακτήρα. Θα ήθελα πραγματικά να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, να ενισχύσουμε την εδαφική διάσταση. Θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο αυτό το σημείο γιατί αυτό παραμένει το βασικό εργαλείο με το οποίο επικοινωνούμε με τους Ευρωπαίους πολίτες. Η εδαφική λοιπόν απόφαση είναι σημαντική. Πώς λοιπόν ενισχύουμε ε, τον ε, ε, εδαφικό χαρακτήρα. Εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και ένα άλλο θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αστική διάσταση έχει ενταχθεί εδώ σε αυτή την πολιτική, αλλά εμείς ασχολούμεθα με την αστική διάσταση που αφορά τις μεγάλες μητροπόλεις. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά μία διάσταση που έχει σχέση με όλη την ε, αστική επικράτεια. το θέμα είναι ακόμα και οι γεωργικές πολιτικές, ε, να δούμε πώς ε, θα μπορούσαν να, ε, να ενσωματωθούν καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεύτερον, το δεύτερο σημείο αφορά το γενικό κανονισμό, αλλά είναι σαφές ότι επηρεάζει και το Περιφερειακό Ταμείο, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλους πόρους. Και αυτό είναι το θέμα της συγχρηματοδότησης και της σχέσης με τη συγχρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σταθερότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί αυτό είναι ένα αποφασιστικό θέμα που καθιστά ακόμα πιο απτά τα προγράμματα. Εμείς προτείνουμε μία ενίσχυση της συγχρηματοδότησης παρόλα αυτά οι περιορισμοί του, ε, της συμφωνίας σταθερότητας μερικές φορές όπως ε, είδαμε και με, από την εμπειρία της Ελλάδας μας έκανε να καταλάβουμε ότι υπήρχαν προβλήματα στη φάση εφαρμογής του προγράμματος. Ενδεχομένως λοιπόν θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο το θέμα αυξάνοντας τις ευθύνες των περιφερειών, όχι αφαιρώντας ευθύνες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για αυτά τα σημεία. Το πρόγραμμα είναι αρκετά φιλόδοξο, θα πρέπει να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο έκθεσης μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να ε, υποβληθούν οι τροπολογίες και τον Νοέμβριο να υποβληθεί στην Επιτροπή. Δηλαδή, στην ουσία μιλάμε για δύο μήνες σκληρής δουλειάς. Αλλά νομίζω ότι και από τις συζητήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες, αλλά και από τη συζήτηση που θα γίνει τώρα στην Επιτροπή, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει μια σωστή δουλειά με την συμμετοχή όλων των συναδέλφων, αλλά και με την βοήθεια της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now... Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης ηγετές, ξεκινώντας με τον κύριο Βαλκάρσελ Σίσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον εισηγητή μας, τον κύριο Κοτσολίνο γιατί όντως η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρκετά θετική. Αλλά, όπως πάντα, υπάρχουν κάποια θέματα που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και συντονισμού. Και γι' αυτό θα συνεργαστούμε για να εμπλουτίσουμε την έκθεση του κ. Κοτσολίνο. Θα προτείνουμε, όπως έκανε και ο εισηγητής, να αναλύσουμε πιο διεξοδικά τα άρθρα 2 και 3 που αφορούν τους ειδικούς στόχους και τη θεματική συγκέντρωση των δύο ταμείων. Και καλό θα ήταν να βρούμε μια ισορροπία ώστε να δώσουμε στις τοπικές και στις περιφερειακές αρχές μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, των δύο ταμείων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πόσο είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε το καθάριστο εγχώριο εισόδημα, κάτι που αναφέρει ε, το άρθρο 3 ως κριτήριο. Στα πλαίσια του γενικού στόχου είμαι υπέρ της συμπερίληψης στο κείμενο κάποιων προβλημάτων που είναι ε, σημαντικά για πολλές περιφέρειες. Για παράδειγμα, το θέμα της γύρες του πληθυσμού ή το ζήτημα της απερίμωσης κάποιων περιφερειών, γιατί πραγματικά έχουμε απερίμωση ή αγροτικών περιοχών ή περιοχών της δυσπρόσιτων Επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στις σημερινές προκλήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο στο κείμενο είτε στους ειδικού στόχους είτε σε άλλα τμήματα του συγκεκριμένου κανονισμού. Επίσης, δεν θεωρώ ότι όλα τα κριτήρια του αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 6 είναι κατάλληλα ή σωστά. Για παράδειγμα, δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Ε, είναι σημαντικές αυτές οι πράξεις ε, ε, και οι ενέργειες αυτές για να προωθήσουμε μια πιο κυκλική οικονομία και πιο βιώσιμη οικονομία. Γιατί να αποκλείονται τέτοιε ενέργειε. Επίση, καλό θα ήταν να συμπεριλάβουμε και άλλε δράσει στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, αλλά και στα κονδύλια που προβλέπουμε για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, κάτι που αναφέρεται στο άρθρο 9. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φίτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο Κοτσολίνο. Επειδή είναι μια πρώτη δυνατότητα Ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που με βρίσκει σύμφωνο και ιδιαίτερα ό,τι αφορά το σημείο εκκίνησης αλλά και σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες του παρελθόντος. Γιατί θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια να επικεντρωθούμε την αποτελεσματικότητα γιατί οι πόροι βεβαίως έχουν συρρυχνωθεί. Τα σημεία που αναφέρθηκαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα ήθελα να διατυπώσω δύο σκέψεις ακολουθώντας το του Το πρώτο σημείο αφορά την διοικητική απλοποίηση. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει, θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης, αλλά θα πρέπει να διορθώσουμε και ορισμένα σημεία. Επιτρέψτε μου να παραθήσω μερικά παραδείγματα που αφορούν την διαχείριση του κάθε ταμείου. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια πώς θα γίνει αυτή η απλοποίηση σε επίπεδο απλού ελέγχου, λογιστικού ε, ελέγχου, σύνδεσης ε, με τις ε, υπάρχουσες τεχνολογίες. Γιατί ο κίνδυνος είναι ότι πολλές φορές χρειάζονται χρόνια για να εφαρμοστούν αυτές οι πρωτοβουλίες και πολλές φορές γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό το πρόγραμμα. Το δεύτερο σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω είναι το θέμα που έγινε παράδοξο της σύνδεσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το να υποστηρίξουμε το θέμα της το είναι ένα θέμα πάρα πολύ σωστό. Το να το θέτουμε ως ε, όρο ε, είναι πραγματικά ένα παράδοξο και υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να υπάρξει ένα σημείο αναφοράς, γιατί μερικές φορές έχουμε διαθέσιμους φόρους, ενώ υπάρχουν αυτοί που μπορούν να κρυφτούν πίσω από αυτό το μηχανισμό για να κρύψουν ε, ατέλειες ε, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλα θέματα. Το νόημα όμως είναι ότι το μήνυμα που στέλνετε είναι ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μία προσπάθεια να κάνουμε μία όσο γίνεται ευρύτερη σύνθεση για να μπορέσει να ε, δοθεί ε, μία εικόνα αξιοπιστίας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού της Πολιτικής Συνοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι η υποφερόμενη Πρόεδρο, ή επόμενη και οδησηγητήρια εκ μέρου των φιλελευθέρων. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω και εγώ λοιπόν κάποιε προκαταρκτικέ σκέψει για την έκθεση Κοτσολίνο. Πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι η πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη και Ταμείου Συνοχής είναι πιο σύντομη και πιο απλουστευμένη με βάση, για τους εφαρμοστέους κανόνες που θα διέπουν και τα δύο ταμεία και χαιρετίζω την πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη φιλοδοξία της να πλουστεύσει τους κανόνες για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Επίσης, επισημαίνω την ανάγκη να καλύψουμε με την πρόταση αυτή όλες τις περιφέρειες, το σύνολο των περιφερειών Έχουμε ένα σταθερό προπολογισμό για το ΕΤΠΑ και έχουμε αύξηση 1%, αλλά ταυτόχρονα στο Ταμείο Συνοχής έχουμε σημαντική μείωση, περίπου 46%. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τον αποδεδειγμένο αντίκτυπο των δράσεων του Ταμείου Συνοχής είναι πραγματικά κρίμα αυτή η μεγάλη μείωση. Χαίρομαι για την μεγαλύτερη ελαστικότητα των νέων στόχων των νέων πέντε στόχων πολιτικής ε, σε σχέση με τις προηγούμενες 11 έχουμε μια μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση και επίσης ε, έχουμε μια καλύτερη επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το πιο κεντρικό κριτήριο ε, το θέμα της θεματικής συγκέντρωσης για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Ταμείο σε, σε, σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, ε, σε επίπεδο δηλαδή ΝΑΤΣ 2. Μεγάλη αλλαγή αυτή η θεματική συγκέντρωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επίσημη υπέρ το 6% για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη ε, σε ό,τι αφορά ε, τα κονδύλια του ΕΤΠΑ για το εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία. Αυτή είναι δεδηλωμένη και επίσης στηρίζουμε τις εξόχως απόκεντρες περιοχές για να αντιμετωπίσουν τις ιδιάζουσες προκλήσεις τους. Η πιθανότητα μεταφοράς μέχρι 5% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στα νέα ε, χρηματοδοτικά μέσα του InvestEU και στα νέα προγράμματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συμβάλλουν στην συμπληρωματικότητα και στην καλύτερη συνέργεια μεταξύ του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και άλλων ε, χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όμως ε, να μεριμνήσουμε τη διαφύλαξη της περιφερειακής διάστασης αυτών των επενδύσεων ε, και την ανάγκη να ληφθούν υπόψη στις εθνικές πρωτοβουλίες. Επίσης, οι δείκτες ε, προσδιορίζονται πολύ καλύτερα σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Με τους καλύτερους δείκτες θα έχουμε και καλύτερη καταμέτρηση ε, της εφαρμογής, του αντικτύπου εφαρμογής και θα βελτιώσουμε την προετοιμασία των προγραμμάτων. Ευχαριστώ τον εισηγητή και περιμένω το σχέδιο εκθεσής του για να ε, μπορέσουμε να υποβάλουμε και τροπολογίες. Παίρνω τώρα στην επόμενη σκιώδη την κυρία Μισελ. Ähm, Ευχαριστώ και εσά κυρία Πρόεδρε καθώς και τον εισηγητή. Θα σύντομη διότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το συζητούμε και θα τονίσω αυτά που θεωρώ ως πιο βασικά προβλήματα. Είμαστε υπέρ της μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευσης. Αυτό ναι, πάντοτε στην παρούσα Επίτροπη θεωρήσαμε ότι αυτό αποτελεί ας πούμε μια εντολή που μας δίνουν και πολλά όργανα περιφερειακά και τοπικά. Και θεωρούμε ωστόσο ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για το ζήτημα της αποκέντρωσης. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μελλοντικά οι προτεραιότητες προώθησης θα συζητούνται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κεντρικές κυβερνήσεις. Γιατί και μάλιστα θα ενισχυθεί αυτό εγώ θεωρώ ότι πρόκειται στην ουσία για παραβίαση της αρχής της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών και ιδίω του τοπικού επίπεδου. Εμείς θέλαμε άλλη κατεύθυνση να λάβει. Κατεύθυνση η οποία θα ενισχύσει το επίπεδο των τοπικών οργάνων. Τοπικό επίπεδο δηλαδή. Ενώ βλέπουμε τώρα ότι οι εθνικές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν πάλι τα ενία. Θεωρούμε ότι αυτό θαμπώνει την εικόνα και θαμπώνει και τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, δεν βλέπουν το ίδιο καλά τις λεπτομέρειες στις εθνικές κυβερνήσεις. Δεύτερο, για την θεματική συγκέντρωση και ιδίως για τις τρεις κατηγορίες της οικονομικής ισχύω του εθνικού επίπεδου. Εκεί το θεωρούμε και αυτό προβληματικό, διότι σημαίνει μεταξύ άλλων ότι κάποιες μεταβατικές περιφέρειες και φτωχότερες περιφέρειες των πλουσιότερων χωρών θα έχουν μόνο στόχους του 3, 3 έως 5. Καλύτερη διαδικτύωση, κοινωνική Ευρώπη και Ευρώπη πλησίων στον πολίτη. Θα δουν εκεί να μειώνονται τα κονδύλια τους για τους στόχους αυτούς. Εκεί θα συμφωνήσω εγώ και με την τάση που βρίσκεται από τη δική μου περιφέρεια του Βερολίνου. το ζήτημα της αστικής διάστασης που στην ουσία θέλαμε να τονώσουμε και να προωθήσουμε. Βλέπω εδώ να τίθεται σε κίνδυνο. Επίσης, πέντε στόχοι. Θα μπορούσα να τους δεχθώ. Θα χρειαστεί και ελπίζω ότι θα επιτευχθεί μια μεγαλύτερη ευελιξία. Όμως, όπως είναι τώρα διατυπωμένοι οι στόχοι πολιτικής, ιδίως ο τέσσερα, κοινωνική Ευρώπη, και τα υποσημεία ε, όπου εμφανίζονται για παράδειγμα η κοινωνική συμπερίληψη, πολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά δεν εμφανίζονται σχεδόν καθόλου τώρα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι το πράγμα. Επίσης, έχουμε μιλήσει για το ζήτημα της επίτευξης των ε, κλιματικών στόχων. Και εδώ είναι πολύ ασαφή τα όσα περιλαμβάνονται. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό περιλαμβάνεται στο διατάφτα, αλλά δεν περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο. Διερωτώ αν θα περιληφθεί στον γενικό κανονισμό. Όπως είπε και ο εισηγητής, έχουμε και εμείς ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με την λίστα των τομέων παρέμβασης που έχουν αποκλειστεί. Για παράδειγμα, επενδύσεις στην στέγη έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θεωρούμε όχι και τόσο καλό, ας το πω έτσι το ίδιο για οχήματα που κινούνται με υγραέριο. Και εδώ νομίζω ότι είναι ασυνεπές αυτό που προτείνεται. Το ίδιο για τις μακροοικονομικές προτεραιότητες, αλλά αυτό το είπα ήδη. Θα αρκεστώ σε αυτά τα σημεία κριτικής για την ώρα. Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε σε συνεργασία με τον εισηγητή και βεβαίως θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρόπε, εσείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, λίγα λεπτά χρειάζομαι μόνο. Είναι σημαντικό να γίνει ανταλλαγή απόψεων τώρα. Να προετοιμαστούμε για τη σύνταξη του κειμένου. Χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται απλούστευση. Σε αυτά συμφωνούμε και είναι και ωραία λόγια. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι ποια πράγματα θα απλουστευθούν και ποιος θα υποφεληθεί από αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι χώρες μέλη. Οι χώρες μέλη ίσως προσφέρουν κάποια χέγγια αλλά το ζήτημα είναι να μην αντιμετωπίσουν περισσότερα εμπόδια οι περιφέρειες. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια πράγματα θα γίνουν αντικείμενα διαχείριση στο συγκεντρωτικό επίπεδο και ποια στο περιφερειακό. Είπαμε ήδη ότι υπάρχουν αλλαγές και μάλιστα πολύ μεγάλες ανάμεσα στι χώρε μέλη. Α μην λησμονούμε ότι υπάρχουν και διαφορές και μέσα στι ίδιε τις χώρε μέλη. Και μιλούμε για μεγάλε διαφορές. Ωστόσο, η χρηματοδότηση θα μειωθεί. Εμείς θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ο ίδιος προϋπολογισμός. Όμως, ακούγεται από παντού το σύνθημα αυτό more for less. Δηλαδή, κάντε όλο και περισσότερα με όλο και λιγότερα χρήματα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι τα όσα είπε ο συγητής είναι σωστά. Θα πρέπει να καθορίσουμε την περιφερειακή διάσταση. Όταν την καθορίσουμε, όταν την ορίσουμε καλύτερα, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για συγχρηματοδότηση. Έχουμε ας πούμε τη συγχρηματοδότηση σε μια πλουσιότερη περιφέρεια, σε μια φτωχότερη περιφέρεια. Θα πρέπει να δούμε τότε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Μίλησε προηγούμενο συναδελφό μου για την ε, υπόθεση του Βερολίνου, για την περίπτωση του Βερολίνου. Υπάρχουν διαφορές, ωστόσο, μεταξύ των περιφερειών, πάρα πολύ μεγάλες. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μα τι σημαίνει εν τέλει περιφερειακή διάσταση και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι περιφέρειες θα επωφεληθούν από τα κονδύλια Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Έχετε άλλα σχόλια, κύριε Βαν Ρόι. Έτοιμα προς τον εισηγητή. Αν κατανόησα καλά τα όσα είπατε, είπατε ότι θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, δηλαδή 8 και 9 Οκτωβρίου. Και είπατε μετά θα υποβάλλετε το σχέδιό σας στις 10 Οκτωβρίου και μετά οι τροπολογίες έχω λίγο μπερδευτεί τώρα με τη διαδικασία, διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην ίδια γραμμή με την CPR. Δηλαδή 27 Σεπτεμβρίου, ήδη το κείμενο προχωρεί στη μετάφραση, μήπως μπορεί να γίνει κάπως πιο αεροδυναμική η διαδικασία αυτή, δηλαδή να προχωρήσει ταχύτερα, να μην έρθει τούτη εδώ έκθεση αργότερα διότι χρειαζόμαστε ταχεία εφαρμογή. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε καθυστερήσει πολύ και ξεκίνησε μετά πάρα πολύ, με πολύ αργό ρυθμό και με καθυστέρηση. Θα απαντήσω εγώ, λέει η Πρόεδρο στην ερώτησή σας, ναι, το χρονοδιάγραμμα είναι να παρουσιαστεί το σχέδιο εκθέσεως στην διάρκεια της συνάντησή μας 8 και 9 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, ξαναλέω θα είναι το σχέδιο εκθέσεως. Τώρα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. 8 και 9 Οκτωβρίου θα είναι περίπου 10 ημέρες μετά από την παρουσίαση του CPR. Την έκθεση, της έκθεσης δηλαδή του CPR. Προσπαθούμε δηλαδή να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες εκθέσεις. Δεν είναι δυνατόν όμως να γίνει στην ίδια συνεδρίαση, διότι πρόκειται για έκτακτες συνεδριάσεις που είναι πολύ σύντομες. Δέκα ημέρε δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, άρα θα είμαστε περίπου εντάξει. Την ίδια ισορροπία θα κρατήσουμε και για τις τροπολογίες. Σας ικανοποιεί η απάντηση αυτή. Βανίστε Ρόι, μπορείτε να μας το δώσετε γραπτός τις ε, προθεσμίες αυτές. Γιάνν Όλμπριχτ. θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τον ε, εισηγητή. Εγώ ετοιμάζω την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού και νομίζω ότι υπάρχουν μερικά αντιφατικά στοιχεία που θα ήταν σκόπιμο να συζητήσουμε. Καταρχάς, αυτό που παρατηρούμε είναι μια αλλαγή στην πολιτική. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή θα, ε, Περιφερειακής θα πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει με την Επιτροπή. Θα θέλαμε να καταλάβουμε ποια είναι η λογική που βρίσκεται από πίσω. Θα πρέπει να γνωρίζει η Περιφερειακή Επιτροπή. Αν έχουμε ένα τεχνητά διεσταλμένο ταμείο ε, συνοχής, αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε αυτή η τεχνητή διαστολή ε, και για ποιο λόγο έχει πάψει να γίνεται αυτή η τεχνητή διαστολή. Δηλαδή, ε, ε, στην ουσία αυτό απευθύνεται στις χώρες συνοχής. Δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα εμπιστοσύνης προς τις χώρες συνοχής. Το Ταμείο συνοχή αφορά τις χώρες συνοχής και αυτό είναι σύμφωνο με τη συνθήκη του Μάστριχ. Νομίζω ότι θα πρέπει το ερώτημα να τύχει μια σαφούς απάντηση Οι άνθρωποι με μας ρωτάνε για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το 40%. Εγώ καταλαβαίνω ότι κινούμεθα προς το φυσιολογικό και μας ρωτάνε για ποιο λόγο. Ε, οι νεοαφιχθέντες ρωτάνε και γιατί δεν ήμασταν φυσιολογικοί. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να ξέρουμε για την ημερησία διάταξη. Γιατί αυτή είναι η Δεύτερη αλλαγή πολιτικής. Η αλλαγή αυτή οδηγεί και σε μια αλλαγή της πολιτικής. Εγώ καταλαβαίνω την κατάσταση μετά την κρίση και τα λοιπά και τα λοιπά. Το αποτελέσμα είναι ότι περισσότερες περιοχές είναι σε φάση μεταβατική. Στη Γαλλία, στη Φιλανδία. Το τρίτο θέμα, πόσα χρήματα θα πάνε στις λιγότερο αναπτυγμένες, στις περισσότερο αναπτυγμένες, αυτές που είναι σε μεταβατική φάση. Τώρα ε, είμαστε στο CPR. Το θέμα ε, αφορά τη συγχρηματοδότηση. Μειώνουμε την ε, συνοχή, αλλάζουμε τη συγχρηματοδότηση, αλλάζουμε την μεταβατική περίοδο, πάρα πολλές αλλαγές. Είναι βέβαια απλοποιημένο αυτό, αλλά εντελώς διαφορετικό. Εγώ δεν τον παραναγαώ αυτό, αλλά θέλω να καταλάβω τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλλαγή των, της ε, θεματολογίας, κέντρωση των σεμάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το έθιξε προηγουμένως και η Επιτροπή. Υπάρχουν δύο στοιχεία, προγραμματισμός και χρήματα σε επίπεδο περιφερειακό. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο εθνικό. Ε, τι εννοούμε όμω λέγοντας κάτι τέτοιο, πολιτικά και γεωγραφικά. Ελπίζουμε ότι θα ε, ε, είναι εδαφικό, αλλά πολιτικά είναι επικίνδυνο. Χρειαζόμαστε και τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή θα γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και θα πρέπει να ακούσουμε και να διαβάσουμε τις παρατηρήσεις των διαφόρων οργανώσεων, CPRM ε, και τα λοιπά. Ποια είναι, αυτή, ποια είναι η αποψή τους για αυτά τα θέματα. Τι συμβαίνει με τα POs, με τα επιχειρησιακά προγράμματα χρειαζόμαστε αυτή τη σοβαρή συζήτηση για το περιεχόμενο. Η πρότασή μου για την Επιτροπή ε, την περιφερειακή πολιτική θα ήταν επικέντρωση σε δύο ομάδες, όχι σε τρεις ομάδες. Θεματική επικέντρωση. Αυτό είναι ένα θέμα εντελώς διαφορετικό. Αλλά αυτή είναι μια λογική. Οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει. Είναι σαν την ε, αστική διάσταση που είπαμε ότι είναι σημαντική. Είπαμε ότι παρατηρούμε μια μετακίνηση σε περισσότερο αστικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο ε, αναφέρθηκα στο θέμα της βιώσιμης ε, αστικής δράσης. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, αλλά χρειαζόμαστε και στην Επιτροπή Προπολογισμού και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη ένα σαφές μήνυμα, το τι συμβαίνει, για ποιο λόγο έχουν επέλθει τόσες αλλαγές, ποια είναι η λογική πίσω από όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους, να τους πούμε ότι εδώ έχουμε αυτή τη διαφορά για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κίλαν. Ε, πραγματικά έχετε δώσει ε, ε, ε, μία παράσταση μόνο σας προσπαθώντας να εξηγήσετε τις αλλαγές. Συμφωνούμε με τις αλλαγές. Μήνες ολόκληρου συζητάμε αυτές τις αλλαγές και αν δεν έχουμε μέχρι τώρα τις απαντήσεις, θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός κινδύνου. Το λόγο, ε, τώρα έχετε πάλι. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Το ίδιο θα έλεγα ότι εδώ και αρκετό καιρό συζητούμε αυτές τις αλλαγές. Οπότε δεν θα χρειαζόταν να, κάνω, να δίνω εγώ παράσταση, να είμαι άνθρωπο ορχήστρα, αν είχε περάσει νωρίτερα το μήνυμα από όλε τι προηγούμενε συζητήσει. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτσολούνα για τι παρατηρήσει αλλά και για την διαλλακτική προσέγγιση του στι συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο κανονισμού. Ήδη είχαμε αρκετά επικοδομητικέ επαφέ και πιστεύω ότι όλοι θα βγούμε κερδισμένοι από το έργο για την πρόθεση του κανονισμού αυτού. Όπως τόνισαν πολλοί ευρωβουλευτές, είναι όντως σύντομος ο κανονισμός, πολύ πιο σύντομος από ό,τι ο προηγούμενος και συνδυάζει την παλιά προσέγγιση των δύο ξεχωριστών κανονισμών για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Και παρόλα αυτά είναι συντομότερο. Αυτό εντάσσεται στη γενικότερη διαδικασία πλούστευσης που προσπαθούμε να πραγματώσουμε και χάρη σε αυτόν τον κανονισμό. Και αυτή είναι η κεντρική απάντηση που θα ήθελα να δώσω στον κύριο Όλμπριχτ, ότι αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο των αλλαγών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ουσιαστική της και αυθεντική της επιθυμία για απλούστευση. Απλούστευση στο περιεχόμενο και την ενάργεια των κανονισμών, απλούστευση για τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και τις αρχές προγραμματισμού που οφείλουν να παρουσιάσουν έργο σε αυτά τα προγράμματα πολιτικής και απλούστευση και για τους δικαιούχους. στη φάση εφαρμογή των επιμέρους προγραμμάτων. Και αυτό βρίσκεται στην καρδιά των προτάσεών μας, η επιθυμία της απλοποίησης. Ε, και αυτό καθοδηγεί όλο το πακέτο των κανονισμών που υποβάλαμε. Και αυτό διέπει όλες τις προτάσεις μας. Στο συγκεκριμένο κανονισμό Προσπαθήσαμε και το τόνισε και ο κύριος Κοτζολίνο να ε, προτείνουμε ένα συνοπτικότερο και σαφέστερο πακέτο για το τι μπορούν να προσφέρουν αυτά τα δύο ε, ταμεία. Γιατί στην τρέχουσα περίοδο έχουμε 11 θεματικούς στόχους, πάνω από 40 επενδυτικές προτεραιότητες και όλα αυτά μπορεί να έχουν νόημα και να είναι χρήσιμα και απαραίτητα για επιμέρους τμήματα και περιοχές της Ένωσης και για επιμέρους προγράμματα, αλλά πώς είναι δυνατόν να το προβάλλουμε σε μια απλή και συνοπτική συνεπιπολιτική Αποκλείεται. Γι' αυτό προτείναμε πέντε βασικούς στόχους πολιτικής και 20 ειδικούς στόχους προσφέροντας έτσι μια πιο συνοπτική προσέγγιση για το πού μπορούν να επενδυθούν τα κονδύλια των δύο ταμείων. Έτσι εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα, προσαρμοστικότητα και δεν χρειάζεται να κατακαιρματίσουμε την χρηματοδότηση σε, πολλά και μικρά πακέτα. Να πω δύο λόγια για τις προτάσεις για τη θεματική συγκέντρωση, γιατί προκάλεσαν έντονα ενδιαφέρον από ό,τι κατάλαβα. Πολύ συχνά άκουσα για τη θεματική συγκέντρωση ε, το φόβο σας για το κίνδυνο να περιορίσει το βαθμό αποκέντρωσης. Θα ήθελα να σας αποσαφηνίσω ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση ε, να συγκεντρώσουμε τη διαχείριση. Καμία προσπάθεια συγκέντρωση δεν κάνουμε γενικώ ούτε στον κανονισμό γενικά, ούτε στη θεματική συγκέντρωση ειδικά. Προτείναμε τη θεματική συγκέντρωση ακριβώς για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο και όχι να μπλοκάρουμε τι περιφέρειες. Κοιτάξτε ένα θεωρητικό παράδειγμα. Με τους υφιστάμενου κανόνες, αν έχουμε ένα κράτο μέλο με δύο περιφέρειες περίπου αντίστοιχου ΑΕΠ, οι δύο αυτές περιφέρειε θα πρέπει να ε, ικανοποιούν ακριβώς τα τις ίδιες απαιτήσει και τις προϋποθέσεις της θεματικής συγκέντρωσης, γιατί γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο αυτά τα κριτήρια. Κάθε περιφέρεια στο πρόγραμμά της θα πρέπει να σέβεται τέτοια ποσοστά. Με την ε, προσέγγιση σε εθνικό επίπεδο έχουμε ξαφνικά μεγαλύτερη ελαστικότητα μεταξύ των δύο περιφερειών. Ναι, μεν θα πρέπει να τηρήσουν τα κριτήρια της θεματικής συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο, και αυτό ευθυγραμμίζεται με τη γενική αρχή της θεματικής συγκέντρωσης, δηλαδή ε, εστιάζουμε τις συνεισφορές των προγραμμάτων μας στις προτεραιότητές μας και γι' αυτό έχουμε ε, τα ε, κριτήρια της θεματικής συγκέντρωσης να εδράζονται στην καινοτομία και στο περιβάλλον. Αλλά σε εθνικό επίπεδο έχουμε ελαστικότητα. Ένα κράτο μέλο που θέλει να ξοδέψει περισσότερα για την καινοτομία μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο της θεματικής συγκέντρωσης γιατί μια άλλη περιφέρεια μπορεί να θέλει να εξοδεύσει λιγότερο για την καινοτομία και περισσότερα στα κοινωνικά θέματα. Στο Βερολίνο, παράδειγμα, θα θέλαμε να επενδύσουν περισσότερο ίσως στην ε, υποδομή, στην κοινωνική υποδομή και όχι στην καινοτομία. Και με τη νέα πρόταση θεματικής συγκέντρωσης επιτρέπεται αυτή η ελαστικότητα. Οπότε είναι πολύ πιο εύκαμπτο και όχι πιο άκαμπτο το σύστημα. Γι' αυτό και προτείναμε τη συγκεκριμένη θεματική συγκέντρωση. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι στο άρθρο 6 έχουμε προβλέψει έναν μακροσκελέστερο κατάλογο από ό,τι στο παρελθόν για τα είδη δράσεις που θεωρούμε ότι εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση των δύο ταμείων. Στόχος μας εδώ είναι να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά. Και εκεί που έχουμε συγκεκριμένη προσέγγιση σε, μια, σε ένα τομέα πολιτικής, περιβάλλον φερρυπίν, ανταγωνισμός ή μεταφορές, θα πρέπει να έχουμε συνεπή προσέγγιση στην παροχή κονδυλίων στις συγκεκριμένες πολιτικές. Εξού και η πρότασή μα για το άρθρο 6 με τις εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχή. Πάντω είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τι συζητήσει και πρόθυμοι και να σας εξηγήσουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία της πρότασής μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κοτσολίνο, θα θέλατε και πάλι το λόγο. Σύντομα παρακαλώ όμως. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανασκουμποθούμε. Να προσπαθήσουμε να δούμε τα θέματα επί των οποίων μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εγώ λέω ότι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και σε ό,τι με αφορά είμαι διατεθειμένος για μια πιο στενή επαφή με τους συναδέλφους ε, προκειμένου να μπορέσει να δοθεί μια απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν εδώ. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γίνει και μια δουλειά προσωμείωσης σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα της θεματικής συγκέντρωσης το θέμα που ετέθη θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάνοντας μία προσομοίωση. Τι συμβαίνει όταν εγκρίνεται ένας νέος ε, κανονισμός. Τι συμβαίνει σε επίπεδο περιφέρειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επισέλθουμε περισσότερο σε θέματα ουσίας. Να είμαστε λιγότερο ασαφείς προκειμένου να καλύψουμε αυτή την ανάγκη από τη στιγμή που υπάρχει ένας απλοποιημένος ε, κανονισμός. Ε, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τα περί πολιτικής ε, συνοχής. Εγώ θα έλεγα αμέσως να ρηχτούμε στη δουλειά και να καταβάλουμε μια προσπάθεια να γίνει μια προσωμείωση που θα μας επιτρέψει να επιλύσουμε προβλήματα και μεταξύ μας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται η ανταλλαγή απόψεων για τη σημαντική αυτή έκθεση. Μένει τώρα ένα θέμα, τα διάφορα. Ένα λεπτό κύριε Βαν Θέμα πρακτικής αξίας. Μέχρι τώρα γνώριζα ότι όταν έρχεται κανείς εδώ, τα πλήρη μέλη έχουν, βρίσκουν στο έδρανό του όλο το πακέτο των εγγράφων. Δεν χρειάζεται να πάνε να τα αναζητήσουν. Τώρα μου είπαν όμως ότι δεν δόθηκε στους ε, ε, κριτήρες της αίθουσας η εντολή να δώσουν το πακέτο των εγγράφων. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Ευχαριστώ, το σημειώνω, λέει η Πρόεδρος. Αν δεν έχετε τίποτε άλλο. Σας παρακαλώ, σας, ε, σας υπενθυμίζω μάλλον ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Στρασβούργο, από τις 10 το πρωί. Αρχίζουμε λοιπόν τις έκτακτες συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ διακόπτεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.